Uh, dear colleagues, can we, can we start the... Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Can we ask them because I don't want to shut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 Dear colleagues, I would like to... Αγαπητοί συνάδελφοι, Λοιπόν, εάν δεν έχετε την κάρτα σας θα ληφθεί υπόψη η ψήφος. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να δούμε αν λειτουργεί ο μηχανισμός ψηφοφοριών. Παρακαλώ να κάνουμε μία δοκιμαστική. Μα καλά δεν έχετε κανένα ψηφίσει. Φαίνεστε όλοι τόσο άπειροι. Ελέγχουμε λοιπόν μία δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Είναι ονομοδότηση, δεν μπορεί να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Εκτό να το ζητήσουν δεν ξέρω πόσοι. Λοιπόν, βλέπουμε 20 κάρτες, αλλά μόνο 17 ψηφίζουν. Δεν ξέρω ποιοι ψηφίζουν επιπλέον. Ο, εντάξει κύριε Κορμπέτ. Λειτουργεί λοιπόν ο μηχανισμός ψηφοφορίας. Πρώτη ψηφοφορία γνωμοδότηση Σιλβί Γκουλάρ για την ε, αναθεώρηση του πλαισίου για την οικονομική διακυβέρνηση έχουν γίνει συμβαστικές προτάσεις και προτείνεται να γίνει από κοινού ψηφορία από την Α μέχρι την J. Συμφωνείτε? Ρίτσαρντ. Θα πρότεινα μία πολύ μικρή προφορική τροπολόγηση στην συμβαστική Α. Να προτείνουμε μόνο δύο λέξεις της εξής. Στη γραμμή 7 της συμβαστικής Α όπου λέει για να διοργανώσουν συγκεκριμένες μορφές διαφοροποίησης και τα λοιπά, Να προσθέσουμε όπου είναι σκόπιμο να διοργανώσουν όπου είναι σκόπιμο συγκεκριμένες μορφές διαφοροποίησης. Ο λόγος είναι προφανής. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καμία διαφοροποίηση. Όταν για παράδειγμα θέτουμε ερωτήματα στον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί αν έχει φορολογικές αρμοδιότητες για παράδειγμα κάποια μέρα η Ευρωζώνη μόνο τα μέλη της Ένωσης που συμβάλλουν σε αυτή τη φορολογική δυνατότητα θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα να ψηφίσουν πρόεδρος. Ωραία. Μα αυτή είναι η καλύτερη διατύπωση. Στους τριμερεί διαλόγους λέμε όπου είναι σκόπιμο λύονται τα προβλήματα. Ωραία, δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τη συμβαστική Α όπως τροποποιήθηκε. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ μισό λεπτό, λέει ο κύριο Γκουαλτιέρη. Τι πάει να πει συνολικά. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Θέλω να υπάρξει κάποια αλλαγή της συμβαστικής K. Ψηφίζουμε για τις συμβαστικές Α, B, C, D, F, I, J. Αυτές, F, I, J. Η A όπως τροποποιήθηκε τώρα από το σχόλιο του Richard Κόμπε. Ποιος είναι υπέρ αυτών των 7 τροπολογιών συμβασμού. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Κανείς. Ωραία. Εγκρίνονται συμβαστική Ή e, όπου E ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της συμβαστικής E, ε. Κατά. Δύο. Άποχες. Μηδέν. Ωραία, εγκρίθηκε και συμβαστική ε. Συμβαστική G. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο κατά. Συμβαστική H όπου έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα της H, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, το δεύτερο τμήμα υπέρ παρακαλώ, κατά Ωραία, ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής H. Α, απέχετε. Δεν πηγαίνετε σε κάποιο άλλο έδρανο, παρακαλώ. Ωραία, άψομα. Λειτουργεί. Λοιπόν, ελέγξαμε και το αποτέλεσμα είναι Απορρίπτεται. 10 υπέρ, 11 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική και να δώσουμε τον λόγο στον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Από ό,τι κατάλαβα θα ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα τελειώνει στη δεύτερη γραμμή με τη λέξη EU. Θα προτείναμε το πρώτο τμήμα να πάει μέχρι την έκτη γραμμή για να καλύψει αυτό το πρώτο τμήμα το οποίο θέλουμε να υπερψηφίσουμε και το σημαντικό σημείο της ισοτιμίας σε κράτος δικαίου και να καλέσουμε η επόμενη έκθεση Φερχόφστατ να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και γι' αυτό παρακαλούμε τις άλλες πολιτικές ομάδες να επανεξετάσουν τη θέση τους έναντι του δεύτερου τμήματος που είναι βραχύτερο και λέει αυτό που θα πρέπει να λέει γενικά, τι δεν πρέπει να γίνεται, να επαγορεύουμε δηλαδή το περιεχόμενο άλλης έκθεσης και πολύ συγκεκριμένα παίρνει θέση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Γιατί αυτό καλύτερα να το εξετάσουμε στην επόμενη έκθεση που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Είμαστε λοιπόν υπέρ ενός ε, μακρύτερου πρώτου τμήματος και γι' αυτό παρακαλούμε να καταψηφιστεί το δεύτερο βραχύτερο τμήμα του, της συμβαστικής ΚΑΠΑ. Ωραία, η πρόταση είναι να μετακινηθεί ο διαχωρισμός των δύο τμήματων. Είστε κατάθετε να μιλήσετε, είστε κατάθετε να μιλήσετε. Γιατί είναι σαν προφορική τροπολογία αυτό. Και τα δύο. Παρακαλώ κύριε Αγκουλά Διαφωνώ γιατί είναι πολύ καθυστερημένη αυτή η πρόταση. Συζητήσαμε επί μακρόν. Ο εκπρόσωπος του, των σοσιαλιστών πάντα εξέφρασε την άποψη της ομάδας του. Δεν θέλω διαδικαστικά κόλπα τελευταία στιγμή, γι' αυτό είμαι κατά. Ο κύριος Γκουαλτιέρη. Βλέπω ότι ο συγητής δεν θέλει να υπερψηφίσει και η ομάδα μας ένα σημαντικό τμήμα της, έκθεσής, ε, της έκθεσής του. Είναι σημαντικό για την ΕΚΟ. τη συνεργασία ε, στο κοινοβούλιο μας, αλλά εντάξει, η εισηγήτρια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πρόεδρος, η γραμματεία μας είπε ότι για κατατμήματα ψηφοφορία μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να υποβληθεί έτοιμα Γουαλτιέρη. Δεν ξέρω αν τεχνικά είναι προφορική τροπολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρόεδρο. Άρα δεν είναι προφορική τροπολογία, αλλά άρα δεν μπορεί να αρνηθούμε το δικαίωμα κατά τμήματα ψηφοφορία, έστω και τελευταία στιγμή. Γκουαλτιέρη. Εντάξει, α το χωρίσουμε σε τρία τμήματα τότε. Το, το πρώτο, δεν θέλουμε, μετά θέλουμε χωριστή ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα, το οποίο επίση θα υπερψηφίσουμε. Οπότε θα μπορούσατε να το δεχτείτε. Πρόεδρος. Σιλβία, ακούσατε την τελευταία πρόταση. Να χωριστεί σε τρία τμήματα. Γουλά Μα το συζητήσαμε εκτεταμένα όλοι οι σκιώδες, το συζητήσαμε. Πολύ θα ήθελα να μου έχουν υποθεί αυτά νωρίτερα. Πρόεδρος. Πέτρο, θες να πεις τίποτα? Όχι. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, η πρόταση αυτή για μία χωριστή κατά τμήματα ψηφοφορία που γίνεται τώρα είναι πάντα στο πνεύμα της διάθεσης συμβασμού που πάντα επιδείξαμε. Ούτως ώστε να επιτευχθούν ευρύτερες συνενέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Α, και ο κύριος Σέπφλιν θέλει το λόγο. Σέπφλιν. Ο Έλμαρ Μπρόκ δυστυχώ ο σκιώδης μας ε, δεν είναι εδώ αλλά όπως είπε η Σιλβί Γκουλάρ έγιναν εκτεταμένες συζητήσεις αυτό είναι το τελικό κείμενο επί του οποίου συμφώνησαν όλες οι ομάδες. Δεν βλέπω να υπάρχουν σοβαροί λόγοι να ανατρέψουμε τη συμφωνία. Οπότε συμφωνώ με την κυρία Γκουλάρ. Πρόεδρος μικρόφωνο. Η κυρία Σπινάλη. Να πω απλώ. ότι δεν κατανοώ, πραγματικά δεν κατανοώ τα επιχειρήματα του κυρίου Γκουαλτιέρη και του κυρίου Περέιρα. Είχαμε όντω πολλέ συναντήσει. και δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί πρέπει να διαρρέσουμε στα δύο και στα τρία τμήματα ένα κείμενο του οποίου εν πάση περιπτώσει είχαμε μια συμφωνία. Συμφωνώ με την κυρία Γκουλά επ' αυτού και εκπλήσωμαι. Εκπλήσωμαι από τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Γιατί βεβαίως πολιτικά υπάρχει υποστήριξη. Γιατί το ΕΛΚ είχε τοποθετηθεί υπέρ της προτάσεώς σας και η το ίδιο είπε. Κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Γκουλάχ, αν υπάρχει υποστήριξη θα ήθελα να είναι πλήρης. Και να μην κρύβονται κάποιοι πίσω από το γεγονό ότι είναι υπέρ της εισαγωγής της οικονομικής διακυβέρνησης ελέγχοντας απλώς ότι ο κύριος Μπερχόφστα δεν τα φροντίσει όλα αυτά. Δηλαδή μπορώ και μόνοι μου να πω ότι εμπιστεύομαι τον κύριο Μπερχόφστα δεν χρειάζεται να το πει η Επιτροπή. Εάν είμαι σε μειοψηφία, καλός. Δημοκράτη είμαι, δεν με ενοχλεί. Ε, την προσέγγιση ψάχνουμε, λέει η Πρόεδρος. Από εκεί και πέρα η ουσία εξαρτάται από τα μέλη. Ε, η κυρία Πέρες. Ευχαριστώ. Είμαστε εν μέσω ψηφοφορία. Είναι κάπως δύσκολο να ξανανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Παραλλήλω, ε, η πρόταση του κύριου Γκουαλτιέρη ε, έχει ως πρόθεση να βελτιώσει την πρόταση. Και εκ μέρους της ε, Οικονομικής και Νομισματικής ε, Επιτροπής νομίζω ότι θα πρέπει η εισηγήτρια να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στο μεγαλύτερο δυνατό τμήμα του κειμένου και αυτό προσπαθεί να κάνει ο κ. Γουαλτιέρη. Άλλοι συνάδελφοι είπαν ότι είχαμε από την αρχή συμφωνία του εδαφείου, αλλά όλοι γνωρίζουν και δεν θέλω να ξανανοίξω τη συζήτηση. Πάντοτε όμως είχαμε πει σε κάθε περίπτωση και ο Πέτρο θα το θυμάται τη βασική μας αρχή και βασική μας θέση από αυτού. Η πρόταση του κυρίου Γκουαλτιέρη που διευρύνει τη στήριξη επί της συμβαστικής προτάσεως που στηρίζουμε είναι καλή την πίστη και θα έπρεπε να είναι καλοδεχούμενη από όλους. Δεν είχαμε συζήτηση από αυτού στην Επιτροπή για τις τροπολογίες αυτές συμβαστικές. Υπάρχουν εξελίξεις τελευταία στιγμής και άλλες ε, ε, υποβλήθηκαν. Όλοι δεχτήκαμε τον κύριο Κόρμπετ ως χρήσιμη πρόταση της τελευταία στιγμής. Ας είμαστε λοιπόν υπαρκώς ε, ευφυείς εστιαζόμενοι στα πράγματα που έχουν σημασία, στα σημαντικά πράγματα έναντι σε μια τροποποίηση της ειδίκης. Δηλαδή. Ελπίζω πραγματικά να είμαστε σε θέση όλοι να προτείνουμε άλλη μια τμηματική ψηφοφορία δηλαδή μια δεύτερη πέραν αυτής που είχε ήδη προταθεί ή και μια τρίτη και δεν χρειάζεται επ' αυτού να περιχαρακωθούμε τώρα όλοι εδώ, νομίζω. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος. Έχω ακόμα δύο μέλη που ζητάνε το λόγο. Ρομπέρτο και Σιλβί, ελπίζω να πλησιάζουμε σε κάποια λύση. Γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Ποιος θέλει πρώτος. Ε, να απαντήσει στην Περβόνς. Όταν διαπραγματευόμαστε με τους κοιόδης, και εγώ πάντοτε αυτό έκανα, εδώ, έχουμε μια κοινή, ένα κοινό όραμα, μια κοινή πρόθεση. Καλώ τα λέει η κυρία Περέζ, αλλά είχαμε μία συνολική συμφωνία επί ενός συνολικού αριθμού συμβαστικών προτάσεων και υπάρχει μία επικονομητική πρόταση που θέλω να σας ε, προτείνω, αν θέλει η ομάδα να με ακολουθήσει. Και μπορούμε να ψηφίσουμε όλοι και είναι ένα πραγματικό βήμα. Τώρα να μην αποδεχόμαστε, δηλαδή να μην παραπέμπουμε στην έκθεση Verhofstadt, που εγώ βρίσκω ότι αλλάζει αλλάζει το, την ισορροπία των συμβασμών που είχαμε επιτύχει, είτε αυτά προερχό... εκφράζονται από τον ΚΟΕ ή από άλλη πολιτική ομάδα, δεν θέλω να τρώω πίσω. Γιατί είναι τσούφε αλέσεις, όπως λέμε. No. Yeah, Τελευταίος ο μιλητής, παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ γρήγορα, λέει ο κ. Γουαλτιέρη. Ο σκιώδης S&D είχε προτείνει τροπολογία, ήταν κατά δηλαδή τη τρίτη θυματική ψηφοφορία. Και είχα ζητήσει και από την Mercedes, για να την αντικαταστήσω, μάλλον είχα πει ότι είναι πρόβλημα. Είναι σημαντικό πρόβλημα σε μια σημαντική γνωμοδότηση και πρέπει να το αποφύγουμε. Για μας είναι σημαντική η ψηφοφορία αυτή. Δηλαδή έχει αντίκτυπο επί του συνόλου της γνωμοδότησης. Όπως είπε και η κυρία Σπινέλη, βρίσκω περίεργο κατόπιν ετήματος σημαντικής αλλαγής που αλλάζει το φάσμα όλης της ε, μελέτης γιατί είχαμε μιλήσει για Eurobond και διάφορα άλλα μιλούν διάφοροι μαζί ομιλητές Γκουαλτιέρη μου, μου ρωτήθηκε, μου υπευλήθη η ερώτηση γιατί αλλάξαμε γιατί τοποθετηθήκαμε έτσι. Το αίτημα ψηφοφορία κατά τμήμα ήταν ακριβώς ένα, μια συμβαστική προσπάθεια. Για να κρατήσουμε τη θέση αυτή στο τελευταίο τμήμα. Είναι ελεύθερη η ψηφοφορία, ο καθένας μπορεί να τοποθετείται όπως επιθυμεί. Αλλά πρέπει να διακρίνομαι. Δεν είναι η στιγμή πράγματι να έχουμε συζήτηση από τη ουσία διαδικαστικά ζητούμε νέα τμηματική ψηφοφορία για να ψηφίσουμε υπέρ στο δεύτερο και κατά στο τρίτο. Κοιτάξτε λέει πρόεδρε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. τελευταίο ομιλητή σίγουρα τώρα. Πρόεδρε, θέλω το εξή να πω στον κύριο Γκουαλτιέρη. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η τροποποίηση συνθήκη δεν έχει διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά στο κείμενο του ΚΕΙ, του μήματος, λέμε μεταξύ άλλων μία από τις προτεραιότητες είναι το κράτος δικαίου κτλ. Είναι τεράλια. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κράτος δικαίου και το δικαστήριο στην τροποποίηση της συνθήκης. Πρόεδρος, κοιτάξτε, έχουμε αποδεχθεί και κανονικά δεν αποδεχόμαστε την ψηφοφορία κατά την τελευταία στιγμή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το επιχείρημα αυτό. Από εκεί πέρα, οι σοσιαλιστές από ό,τι κατάλαβα θα ήθελαν ε, ένα ευρύτερο τμήμα να έχουν για να μπορέσουν να υπερψηφίσουν και να μειώσουν αν θέλετε την καταψήφιση μόνο στο τελευταίο τμήμα. Είναι καλή πρόθεση αυτό, είναι καλή πίστη. Γνωρίζω ότι είναι σημαντικό θέμα. Αλλά εδώ οι σοσιαλιστές έχουν το δικαίωμα να το ζητήσουν έτσι. Ζητώ λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία από των τριών τμήματων του ΚΕΙ από το belief στο πρώτο τμήμα μέχρι την TU. Δεύτερο από το considers μέχρι το European Union και τρίτο τμήμα είναι το υπόλοιπο. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της συμβαστικής και παρακαλώ. Sorry. Yes, I, I, I can try. Μπορούμε να προσπαθήσουμε αυτό. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε αργά, ξανά, πώς θα χωρίσουμε το δεύτερο τμήμα. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα στη δεύτερη αράδα. Το TEU, μέχρι εκεί. Έπειτα αρχίζει το δεύτερο μέρος, το οποίο τελειώνει στην έκτη αράδα με τη λέξη European Union. Το βρήκατε? Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρας. 19 ψήφοι υπέρ, μία κατά, δύο εποχές. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα, από το Considers μέχρι το Union. Πέρας. 19 υπέρ, μία κατά, δύο κατά. Και πάμε τώρα στο επόμενο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν 13 υπέρ 9 κατά. Καμία αποχή. Εκτός μικροφώνου πρόεδρος. Μάρκος Πρέτσελ, τροπολογία είναι. Ποιος είναι υπέρ. Νομίζω πρέπει να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά γιατί μισή από εσά δεν σηκώσατε το χέρι σας. Ή ήσασταν κατά. Λοιπόν, ποιο είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, σαφέστατα. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά μπορούμε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με 5 ψήφους υπέρ 16 κατά. Ε, νομίζω πως υπάρχει ένα μικρό λάθος στον κατάλογο ψηφοφορία, στον κατάλογο των εισηγητών. Γιατί υπήρχε ένα συν, δεν ξέρω γιατί βλέπω τώρα. Συν, υπήρχε πλήν μάλλον. Ναι, και εγώ συν έχω. Η τροπολογία 14 καλύπτεται μόνο εν μέρη από τον συμβιβασμό A, γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσουμε τώρα το υπόλοιπο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ? Ποιος είναι κατά? ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 14. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Με 9 ναι, υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 16. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Η οποία καλύπτει μόνο ένα μέρος από τον συμβασμό F. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 27 αποσύρεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και η 34 ερωτηματικά ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Σωστά. Βέβαια, απορρίπτεται. 35. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται. Αλλά μπορούμε και να επαληθεύσουμε. Καλύτερα. Τροπολογία 35. Πέρας. Απορρίπτεται. Με 13 ψήφους κατά και 8 υπέρ. Τροπολογία 36 και αυτή μέρος του συμβασμού 1. Ε, άι, ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 36. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. Ναι, απορρίπτεται. Τελειώσαμε λοιπόν. Τελική ψηφοφορία. Είναι μια γνωμοδότηση, οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αν το επιθυμείτε όμως, ας το κάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν με 12 ψήφου υπέρ, 3 κατά και 7 αποχές. Εγκρίθηκε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Περνάμε τώρα σε άλλη μια ψηφοφορία για την ερμηνεία του εσωτερικού κανονισμού. Μας ζητήθηκε από την Επιτροπή Γιούρη στα πλαίσια των ακράωσεων των Επιτρόπων να γνωμοδοτήσουμε. Υπήρξε θέμα σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών συμφερόντων, της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Μα ζητήθηκε λοιπόν από την Επιτροπή Γιούρη, από την Ομάδα Εργασίας για τον Εσωτερικό Κανονισμό και θα ήθελα να Απευθύνω το λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Ρίτσαρντ Κόρμπετ, τον επικεφαλής της ομάδας εργασίας, για να μας εξηγήσει γιατί τοποθετήθηκε η ομάδα του με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Να τονίσω ότι αυτή είναι μια ερμηνεία του υφιστάμενου κανόνα του εσωτερικού κανονισμού. Έτσι δηλαδή πώς είναι τα πράγματα τώρα. Με επιφύλαξη λοιπόν για τη διαδικασία κρόαση των επιτρόπων. Αναφέρομαι στο αν θα χρειαστεί να αλλάξουμε στο μέλλον αυτόν τον κανόνα. Εδώ αναφέρεται μόνο το τι σημαίνει ο υφιστάμενος κανόνας, δηλαδή πώς εμπλέκεται η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στην αξιολόγηση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των υποψήφιων επιτρόπων, τις οποίες πρέπει να συμπληρώσουν πριν τις ακροάσεις τους. Αναφέρεται λοιπόν ότι όπως έχουν τα πράγματα η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πρέπει να επαληθέσει ότι έχει συμπληρωθεί η δήλωση οικονομικών συμφερόντων φυσικά όχι μόνο για λόγους γραφειοκρατίας αλλά για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων από το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής. Επίσης, η Επιτροπή αυτή είναι η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την ακρόαση θα κληθεί να αποφασίσει πώς θα συνεχίσει. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει διευκρίνηση των υφιστάμενων κανόνων για το πώς θα πρέπει να αλλάξουν σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μια ακρόαση τους επόμενους μήνες. Εάν για παράδειγμα παρετηθεί κάποιος επίτροπος προτού εμείς καταφέρουμε να επαναξιολογήσουμε τον εσωτερικό κανονισμό υπήρξε μια περίπτωση όπου ο Έλληνας Επίτροπος ε, είχε προταθεί για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γι' αυτό αναφέρουμε. Ποτέ δεν ξέρουμε λοιπόν πότε ενδέχεται να φύγει κάποιος Επίτροπος. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να υπάρχει σαφήνεια. Να πω όμως ότι παρόλα αυτά έχουμε τη δυνατότητα τροποποίησης των κανόνων σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας για τις ακροάσεις των Επιτρόπων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πασκάλ Ντουράν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Με ενοχλεί λιγάκι η ανάλυση που μόλις έκανε ο κύριος Κόμπετς. Γιατί έχω εντελώς αντίθετη άποψη. Όχι επί της ουσίας, αλλά επί των διαδικαστικών λεπτομεριών. Γι' αυτό θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε και να αναβάλουμε την ε, ψήφιση για το θέμα αυτό. Γιατί αυτή η ερμηνεία στην ουσία τροποποιεί τους κανόνες. Τα κείμενα είναι σαφέστατα. Η ζουρή πρέπει να εξετάσει αν και κατά πόσο είναι αποδεκτή μια δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Αυτή την εξέταση την κάνει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Αυτή τη στιγμή οι επιτροπές που κάνουν τις ακροάσεις εξετάζουν μόνο το θέμα των ικανοτήτων του υποψηφίου επιτρόπου. Κατά πόσο είναι κατάλληλος. Προς τη στιγμή η ζουρή απλώς έλεγχε εάν ήταν σωστά συμπληρωμένη η δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Είναι πρόοδος αυτό, συμφωνώ. Αλλά πιστεύω ότι για να είμαστε συνεπείς θα έπρεπε η ζουρή στα πλαίσια των ε, συμφωνημένων κειμένων και συνθήκων εξετάζει εάν ή όχι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων γιατί αυτό είναι το θέμα της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων εάν προκύπτει από αυτή τη δήλωση σύγκρουση συμφερόντων και γι' αυτό πρέπει να τεθούν ενδεχομένω συμπληρωματικέ ερωτήσει και οι αρμόδιε επί τη ουσία επιτροπέ εντό των συνθηκών ελέγχουν εάν έχει τι αναγκαίε ικανότητε. Αυτό που προτείνεται τώρα, που το καταλαβαίνω, είναι το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων, που είναι νομικό θέμα, να το θέσετε στο ίδιο επίπεδο με την καταλληλότητα, που είναι ένα πολιτικό θέμα τεχνικοπολιτική αλλά κυρίως πολιτική. Εάν συμφωνείτε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, να το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω, γιατί έχω την εντύπωση, αν ψηφίσουμε τώρα, παραβιάζουμε τις συνθήκες και ε, θα υπάρξουν επιπτώσεις. Επί της ουσίας ε, δεν νομίζω ότι διαφέρουμε τόσο πολύ. Πρόεδρος. Οι συντονιστές ζήτησαν να το συζητήσει η ομάδα εργασίας. Στην ομάδα εργασίας συζητήθηκε και η δική σας άποψη. Αλλά η ομάδα εργασίας πρότεινε, λαμβάνοντας υπόψη την αντίθεσή σας, να ψηφίσουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε, παρά το έτοιμά σας κύριε Ντουιρό. Ή μπορούμε, εάν η πλειοψηφία το θέλει, να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Αλλά δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε τη διαδικασία που όλοι θέλαμε, που ήταν να περάσουμε ομάδα εργασία η οποία να προτείνει μια λύση. Τώρα πρέπει να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε αυτή τη λύση. Οπότε προτείνω να ψηφίσουμε. Αλλά έχει υποβληθεί διαδικαστικό αίτημα να αναβληθεί η ψηφοφορία. Δεν ξέρω τώρα θα αλλάξει τίποτα. Γιατί η ομάδα εργασία έκανε την πρότασή του. Την πρότασή τη και είναι σεφέστατη. Ο Ρίτσορντ. Αφού δεν θέλετε να μπούμε στην ουσία, καλώς. Καλώς. Γιατί επί της ουσίας διαφωνώ με την ανάλυση, αλλά αφού δεν μπορώ να διαφωνήσω δεν θα πω τίποτα. Αλλά το συζητήσαμε στην ομάδα εργασίας για τους κανόνες, το είπα, και το κρίναμε ομόφωνα νομίζω. Στα όλες οι πολιτικές ομάδες θεωρούσαν ότι αυτή ήταν ικανοποιητική λύση. Ερμηνεύοντας τον υπάρχοντα κανόνα, χωρίς να αποκλείουμε μεταγενέστερη τροποποίησή του. Θα συζητήσω μετά με τον κύριο Ντιρόν γιατί νομίζω ότι δεν συμφωνώ με την ανάλυση του επί της ουσίας. Πρόεδρος. Μα αυτή είναι η διαδικασία που επιλέξαμε. Τώρα η Επιτροπή μας πρέπει να, να ψηφίσει την πρόταση που μας έρχεται από την ομάδα εργασίας. Οπότε να περάσουμε στην ψηφοφορία που νομίζω ότι πρέπει να είναι ηλεκτρονική. Δεν είναι ονομαστική. Αλλά για να μην χρειαστεί να μετράμε, παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ποιοι είναι υπέρ της ερμηνείας που κάνει η ομάδα εργασίας για το τι εξετάζει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Με απλή πλειοψηφία περνάει. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Θα επανέλθουμε στη ζήτηση αυτών των θεμάτων, γιατί συζητάμε τώρα την αλλαγή του κανονισμού, του εσωτερικού κανονισμού. Δεν αποκλείεται λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση. Ούτως ώστε να συζητάμε διαφορετικά ε, το κατά πόσο είναι κατάλληλος ένας υποψήφιο επίτροπος. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Τη μερική διατάξη τώρα τώρα που τελείωσαν ψηφοφορίε. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. I, we, George, I think we, we wait till they move. Ε, Γιώργη, περίμενα να βγουν παρακαλώ. Όσοι θέλουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα. Η έκθεση του Γιώργη Σέρφλιν για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσοι έχετε παρακολουθήσει το ζήτημα, θα γνωρίζετε ότι το ECI, η Πρωτοβουλία Πολιτών, Είναι ένα κέρια σημασία ζήτημα, διακόπτει ο μιλητή. Okay, so I'll begin again. Of course not. Να ξαναρχίσω, Πρόεδρε. Δεν πειράζει. Ας το, ξαναπώ. Και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ. Όσοι λοιπόν παρακολουθείτε την εξέλιξη του πράγματος, θα γνωρίζετε ότι οι πρωτοβουλίες ε, πολιτών είναι κέρια σημασίας. Έχουμε ήδη δύο φορές αν θυμάμαι καλά ασχοληθεί. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να ενέχονται οι πολίτες με αρκετά άμεσο έμπαστος ή ανάλογα άμεσο τρόπο στα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία τη νομική, την πολιτική ε, σχηματίζοντας γέφυρες, συνδέσμους Άμεση επικοινωνία με του πολίτες και κάτι που θεωρούμε εκπληκτικό, νομοθετικέ πρωτοβουλίε που μπορούν να προέλθουν από κάτω, από το λαό. Και μια δυνατότητα που εμπίπτει στη συνθήκη. Το μέσο αυτό ετέθη ισχύ 1η Απριλίου 2012, δηλαδή έχει λειτουργήσει τρία έτη. Και τα όσα επιτυχεί, έχει επιτύχει τα τρία αυτά έτη είναι αρκετά λίγα. Νομίζω 50 ή 51 πρωτοβουλίες. Υπευλήθησαν και δεν έγινε τίποτα ιδιαίτερο με αυτές. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε προβλήματα προκειμένου να λειτουργήσει το μέσο. Μερικές φορές από το περίπλοκο και αντιφατικό πεδίο διάδρασης μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών εθνόντων. Προσπαθώντας να καταλάβω λοιπόν τι συμβαίνει, είχα εκτεταμένες επαφές και διαβουλεύσεις με διάφορους ενδιαφέρομενους φορείς. Θα θυμάστε την ακρόαση που είχαμε 26 Φεβρουαρίου που ήταν πολύ σημαντική και πολύ χρήσιμη. Υπογράμμισε διάφορες πτυχές που δεν τις είχαμε σκεφτεί αρκετοί από εμά. Και στις επαφές λοιπόν που είχα και σε εκείνη τη συνάντηση είχαμε κάποιες προκατακτικές προτάσεις προκειμένου το μέσο αυτό να γίνει πιο εύκολο για το χρήστη και στην ουσία πιο αποτελεσματικό, πιο βιώσιμο. Καταρχά λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα ενδεχομένω ρητορικό. Αυτή τη στιγμή ένα έτος χρειάζεται για τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Ε, έχει υποθεί ότι ενδεχομένω θα πρέπει να γίνει η προθεσμία αυτή 18 μήνες ή και περισσότερο. Τώρα το εκατομμύριο υπογραφών από 7 κράτη-μέλη, το 7 ως τέτοιο, δεν θέτει πρόβλημα εφόσον προφανώς είναι 28 τα κράτη-μέλη συνολικά, αλλά το 1 εκατομμύριο των υπογραφών ερμηνεύεται ως υπερβολικά περιοριστικό. Και ίσως η Κομισιόν εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί μια ευελιξία, δηλαδή αν είμαστε σαφώς πάνω από 900.000, ή τελευταίες δεκάδες χιλιάδων ίσως να μην είναι και τόσο σημαντικές, δεν αλλάζουν και τόσο πολύ τα πράγματα. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι η ιστοσελίδα που αυτή τη στιγμή υφίσταται καλύπτει όλες τις ε, ενδεχόμενες πιθανότητες. Πρέπει πάντως να τη δούμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι φιλική προς το χρήστη. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και γνωρίζω ότι υπάρχει η δημοσιονομική επίπτωση να έχουμε ένα, μια υπηρεσία, ένα γραφείο που να ασχολείται σε κάθε κράτος μέλος με αυτές τις πρωτοβουλίες προκειμένου να βοηθά τους πολίτες να κατανοούν τι δυνατότητες έχουν. Όλα αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα όπως έλεγα και νομικός και τεχνικός και πολιτικός. Μία λοιπόν υπηρεσία που θα μπορούσε να βοηθά. Λέγοντας, ενημερώνοντας πολίτες, ναι αυτό έχει δυνατότητες ή αυτό δεν μας φαίνεται πολύ πιθανό, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό, μην ασχολείστε άλλο. Και νομίζω ότι πριν από τρία χρόνια το είχαμε συζητήσει αυτό. Δηλαδή αν κάποιος προσέρχεται με ένα ECI για την επανεισαγωγή της αναντικής μηνής, ε, κάποιος θα του έλεγε από την αρχή μην το σκέφτεσαι καν, άστο. Βεβαίως και θα υπάρχουν φαιές ζώνες και αμφισημίες που τέτοια βοήθεια θα ήταν πολύ χρήσιμη. Επίσης στη συνάντηση προέκυψε η η πολιτική, αν θέλετε, αποτελεσματικότητα των διοργανωτών και βιωσιμότητα. Και η ευθύνη, η νομική ευθύνη, η οποία θα πρέπει ή να έρθει ή να περιοριστεί σημαντικά. Τώρα η εγγραφή, η καταχώρηση μάλλον, οι κανόνες για την καταχώρηση της υπογραφής είναι 28 και τα κράτη-μέλη. Μερικές χώρες δεν έχουν κανένα σύστημα ταυτοποίησης, άλλες χώρες έχουν αριθμούς, στην Ουγγαρία πρέπει να ε, ε, παράσχει κανείς το μητρικό το όνομα της, το, μάλλον το πατρικό όνομα της μητέρας του, δεν ξέρω γιατί. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μια ομοιομορφία ε, των κανόνων αυτών και η δική μου προσωπική άποψη που την είχα πει στην συνάντηση είναι να κινηθούμε προς ένα ψηφιακό επίπεδο για τους Ευρωπαίους πολίτες, παράλληλα προς την ψηφιακή ατζέντα. Προφανώς δεν θα γίνει εν μία νυχτή, θα χρειαστεί χρόνο, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά και αρκετά σύντομα. Και αυτό άπτεται και άλλων θεματικών που συζητήσαμε το πρωί για την ψηφιακή ψηφοφορία κτλ. Και ότι βεβαίως αυτό δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, αλλά θα έπρεπε να είναι μια δυνατότητα που θα δίνεται εθελοντικός. Ή στην πολιτική διάσταση θέλω να πω ότι το Μισιόν καλό θα ήταν να είναι πιο ανοιχτή. Γιατί βέβαια το ιστορικό τα λέει όλα. Από 51, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει καμία, δεν, έχει, δεν έχουμε καταλήξει σε καμία νομοθετική πρόταση. Έχει γίνει δεκτό το δικαίωμα το δικαίωμα ως αρχή για το νερό, αλλά δεν έχει οδηγήσει σε κάποιο αυτό νομοθέτημα η πρόταση. Ε, δεν, δεν ξέρω αν εκκρεμεί κάτι στο δικαστήριο. Είχαμε μιλήσει για την ανάγκη ακροάσεων συναντήσεων πριν, τις, πριν την εκκίνηση των πρωτοβουλειών, το είχαμε πει στο Κοινοβούλιο και υπάρχει και μια κατάσταση όπου τα νομικά θέματα και οι πολιτικοί ηθήνοντες συναντώνται ε, και αυτό είναι το άβολο. Η Κομισιόν ε, έχει ε, ορίζει τους κανόνες, αποφασίζει μόνη της, απορρίπτει. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα έπρεπε να εισαχθεί κάποιο είδους σύστημα διατησίας ή επίλυσης διαφορών, εν πάση περιπτώσει προκειμένου να γνωρίζουμε τι είναι απορριπταίο και τι όχι. Ελπίζω να λάβω καινοτόμε προτάσεις από τα μέλη. Ευχαριστώ πολύ, Κιόρκη. Ο Γιολάινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και Εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ η ακρόαση, γιατί πραγματικά ήταν πλουσιότατη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Να, και μάθαμε πάρα πολλά για τη διαδικασία στην πράξη. Πάρα πολλές ε, κυβερνήσεις πιστεύω υποτίμησαν την ε, αξία της διαδικασίας ακροάσεων και τώρα έχουμε περάσει στην άλλη πλευρά ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες πολιτών είναι επιτυχείς. Ο Γιώργης να ανέφερε πάρα πολλά σημαντικά θέματα αυτό το διάστημα των 12 ή 18 μηνών πιστεύω πως ε, πρέπει να το σκεφτούμε. Έπειτα το 1 εκατομμύριο υπογραφές ε, να πω ότι βρίσκεται στις συνθήκες και πρέπει να τις πάρουμε στα σοβαρά. Εντάξει, υπάρχει ίσως διαφορά ανάμεσα σε 940.000 και 980.000 υπογραφές, όμως το όριο είναι ένα εκατομμύριο υπογραφές και αυτό είναι κάτι σαν κόκκινο φανάρι. Εντάξει, δεν ε, είναι λίγο ή πολύ κόκκινο, όταν είναι κόκκινο είναι κόκκινο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να παίζουμε με τον αριθμό των υπογραφών που χρειάζονται. Επίσης, από την ακρόαση κατάλαβα την ουσιαστική διάσταση της πρωτοβουλίας των πολιτών και αν η αρμοδιότητα εμπίπτει στην Επιτροπή ή αν είναι στα πλαίσια των συνθήκων. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ο κύριος Σόπφλη να πει κάτι από αυτού. Εάν δηλαδή περιορίζονται οι πρωτοβουλίες αυτές ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εάν όχι. Επίσης, διατυπώθηκε το ερώτημα του αν αυτές οι πρωτοβουλίες απευθύνονται μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι στο Συμβούλιο ή και στο Κοινοβούλιο. Κατά τα άλλα πιστεύω πως οι προτάσεις είναι πάρα πολύ καλές και θα πρέπει να τις στηρίξουμε και να δημιουργήσουμε λοιπόν μία υπηρεσία, ένα γραφείο στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες, ε, ένα γραφείο σε κάθε κράτο μέλο, κράτος μέλος ίσως, διότι ένα ε, πράγμα για το οποίο μας κατηγορούν είναι ότι δεν ενημερώνονται επαρκώς οι ετώντας για την εξέλιξη της αίτησής τους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σιλβί Κάουφμαν έχει το λόγο για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τον εισηγητή και να πω ότι πραγματικά η ακρόαση αυτή για μένα ήταν ιδιαίτερα σημαντική διότι είχαμε αρκετούς καλεσμένους, διαφοροποιημένους με διαφορετικές εμπειρίες που είχε φέρει ο καθένας στην ακρόαση. Και πραγματικά πιστεύω ότι αντίθετα με άλλες ακροάσεις η συγκεκριμένη ήταν αναγκαία. Γιατί μάθαμε πάρα πολλά. Έχω ένα ερώτημα προς τον ε, εισηγητή. Δεν γνωρίζω μέχρι τώρα εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει πότε θα υποβάλει κάποια σχετική αίτηση Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να την υποβάλει μέχρι την 1η ε, Απριλίου, διότι τότε θα έχει περάσει η προθεσμία των τριών ετών. Δεν γνωρίζω την ακριβή ημερομηνία, αλλά θα με ενδιαφέρε πολύ να μάθω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Εντάξει, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει ότι θα κάνουμε τη μία ή την άλλη τεχνική προσαρμογή στη διαδικασία αλλά υπάρχει και ενδεχόμενο να χρειάζεται να αλλάξει ο ίδιος ο κανονισμός. Και η εντύπωση που αποκόμισα εγώ από την τελευταία ακρόαση είναι ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται όσο έχει. Και πρέπει αυτό το σύστημα της πρωτοβουλίας των πολιτών να αλλάξει και να γίνει βιώσιμο και πιο αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, το χρονοδιάγραμμα συγκέντρωσης υπογραφών. Εσείς λέτε ότι οι 12 μήνες αρκούν, άλλοι λένε ότι 18 μήνες είναι καλύτεροι. Πιστεύω πως για όλους είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει μία αυτοματοποίηση σε αυτό το ζήτημα. Όταν δηλαδή καταγράφεται μία τέτοια πρωτοβουλία, να αρχίσει να τρέχει αυτόματα η προθεσμία συγκέντρωση υπογραφών. Εδώ υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις όπου λένε ότι χρειάζεται να περιμένουμε ένα μήνα μετά την ε, καταγραφή, δύο μήνες έτσι ώστε να μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι διοργανωτές για να αρχίσουν να συλλέγουν τις υπογραφές. Όμως πολλοί από την άλλη οι διοργανωτές λένε ότι δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει με την ε, καταχώρηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να διοργανώσουμε την ε, συλλογή υπογραφών και έτσι γίνεται παράταση και έτσι υπάρχει η καθυστέρηση και έτσι τελειώνουν και οι 12 μήνες πριν προλάβουμε να το καταλάβουμε. Και πιστεύω πως αυτό το ζήτημα ε, της διαδικασίας δηλαδή είναι πιο σημαντικό ίσως από το αν η προσθεσμία θα πρέπει να είναι 12 μήνες ή 18. Επίσης, ο κύριος Σόπφλεν ανέφερε και άλλα ενδιαφέροντα σημεία στην έκθεσή του, για παράδειγμα τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την δημιουργία ενός ε, γραφείου στα κρατη το οποίο δεν θα δίνει μόνο πληροφορίες, αλλά θα παρέχει και νομικές συμβουλές. Και το λέω αυτό διότι έχουμε παρατηρήσει ότι περίπου 40% των ε, πρωτοβουλειών των πολιτών αξιολογούνται μη, ως ε, μη παραδεκτές. Επομένως είναι πολύ δύσκολο ένας πολίτης να μπορεί μόνος του να κρίνει εάν μπορεί να κάνει κάτι ή όχι, από νομική άποψη. Και πολλές φορές όταν λαμβάνει την απόρριψη απογοητεύεται. Και αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους πολίτες παρέχοντας νομικές συμβουλές. Τέλος, πρωτού μακρηγορήσω, να πω ότι σίγουρα θα χρειαστεί να το συζητήσουμε παραπάνω, αλλά θα ήθελα επίσης να συζητηθεί και το θέμα της ηλικία. Ακούσαμε και νωρίτερα σήμερα για το ενιαίο ευρωπαϊκό δικαίωμα ψήφου. Ξέρουμε ότι στην Αυστρία ψηφίζουν από τα 16, αλλά σε άλλα κράτη-μέλη από τα 18. Και οφείλω να πω ότι αυτό δεν το βρίσκω σωστό, διότι πρόκειται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εδώ οι πολίτες θα μπορούσαν να αναλάβουν μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να δρομολογηθεί αλλαγή σε αυτό το θέμα. Να παροτρύνουν την Επιτροπή να κάνει κάτι, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Διότι πιστεύω ότι όλοι οι 16χρονοι και οι 16χρονες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα ψήφου εφόσον σε μία από αυτές θεωρούνται υπεύθυνοι πολίτες. Και πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη που, έχουμε που έχουν οι πολίτες μας σε εμάς και να αναγνωρίσουμε την υπευθυνότητά τους. Και τέλος, απευθυνόμενοι στον εισηγητή, ε, μας αναφέρατε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την εκθεσή σας. Θα θέλατε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, ε, τι γίνεται και στη συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών ε, σχετικά με τις προθεσμίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάιτε Παγκάθα Ουρτουντούα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Γκέρας ε, αλλά η ακρόαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και δεν είναι λεπτομέρεια ένα εκατομμύριο υπογραφέ. Είναι σοβαρό θέμα. Διότι αυτή η πρωτοβουλία δεν πρέπει να είναι αγώνας μετεμποδίων κατά των πολιτών. Εάν οι πολίτες ξεκινάνε μια τόσο φιλόδοξη πρωτοβουλία, εμείς πρέπει να τους διευκολύνουμε να τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν. Εάν ε, και τέτοιες, ε, να μπορούν να αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες, αλλιώς ε, είναι αυτογκόλ. Πέρα όμως από την ε, εισαγωγή ψηφιακών μεθόδων που πρέπει να μελετήσουμε που λέει ο και που θα μπορούσε να βοηθήσει, το θέμα τίθεται το θέμα της απλότητας, ε, της ομοιομορφίας και της διευκόλυνσης των πολιτών. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν αρκετή βοήθεια, αρκετές συμβουλές για να ξέρουν τι μπορεί να είναι αντικείμενο μια τέτοια πρωτοβουλία για να μην υπάρχει αυτή η απογοήτευση. Για να μην υπάρξει απόρριψη των θεσμικών οργάνων γιατί θεωρούν ότι προτείνουν δυνατότητες που τελικά οι πολίτε δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία προσαρμογής και βελτίωση των ε, μεθόδων τώρα και σίγουρα ο κύριο Σόπφλιν θα λάβει όλη μα τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Η Μπάρβαρα Σπινέλη. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, τους συναδέλφους Σότκεμ και Κόφμαν για τις προτάσεις ε, αλλαγών, τροποποιήσεων, μεταρρυθμίσεων προτείνουν και συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω το σημαντικό κίνδυνο να λησμονήσουν, να αγνοήσουν τελείως οι πολίτες ένα τέτοιο μέσο, μια τέτοια δυνατότητα που τους δίνεται. Να θεωρήσουν ότι δεν έχει καμία σημασία και ότι εμείς δεν του δίνουμε καμία σημασία και αυτό πρέπει να το πούμε σαφώς. Η ευθύνη της Κομισιόν είναι συγκεκριμένη. Είχαμε τρεις πρωτοβουλίες πολιτών που έφτασαν στο όριο και πολύ πέραν αυτού του ενός εκατομμυρίου υπογραφών και δεν έγινε καμία παρακολούθηση μετά, δεν έγινε τίποτε άλλο. Δηλαδή ακόμα και όταν καταφέρνεις να φτάσεις στο τέρμα, πάλι δεν γίνεται τίποτα. 20, το 40% δηλαδή απερίφθησαν από την Κομισιόν και αν θυμάμαι καλά, δεν απερίφθησαν όλες λόγω πλαισίου αρμοδιότητας απερίφθησαν ακόμα και μερικές χωρίς να είναι καν σαφές σε ποιον εμπίπτει ποια αρμοδιότητα κτλ. Δηλαδή αφενός δεν υπάρχει καμία παρακολούθηση, αφεντέρου υπάρχει 40% απόρριψη. Και η κυρία Κάφμαν τα περιέγραψε πολύ σωστά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου ομοιόμορφοι οι κανόνες της ε, συλλογής των υπογραφών το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και επιφυλάσσομαι να υποβάλω ένα προμεμόρια επί του θέματος αυτού για μια συνάντηση που έχω διοργανώσει αύριο μαζί με τον Κάστενμπεργκ ε, και ίσως να είναι ε, χρήσιμο για την Επιτροπή θεσμικών υποθέσεων να γνωρίζει και τα πορίσματα αυτής της συνάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ λέει πρόεδρο. Ο κύριο Κόρμπετ είναι ο τελευταίο ομιλητή του κατάλογό μου. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα γνωρίζετε ότι πάντα είχα μια άποψη δεν θαύμαζα ποτέ ιδιαίτερα πολύ την το μέσον αυτό, το θεσμό αυτόν έτσι όπως είχε αναπτυχθεί. Είχαμε μια καλή ιδέα που ήταν υποβάλλουμε στην Κομισιόν και η Κομισιόν ίσως να συμφωνήσει αν έχετε ένα εκατομμύριο υπογραφής και αν καταχωρήσετε και το πατρικό όνομα της μητέρας σας ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο εντός στενής ε, χρονικής προθεσμίας ώστε να δυσκολεύεστε ακόμα περισσότερο είναι παλαβό. Δηλαδή οποιοδήποτε θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα, εφόσον έχει μια καλή ιδέα, να την υποβάλει στην Κομισιόν και η Κομισιόν να λάβει δράση. Όμω, το πράγμα είναι στη συνθήκη, ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο λιγότερο γραφειοκρατικό γίνεται, μπα και λειτουργήσει. ώστε να ανταποκρίνεται η Κομισιόν όταν λαμβάνει εν πάση περιπτώσει μία πρωτοβουλία που δείχνει να μπορεί να έχει τόσο ευρεία συνένεση μεταξύ των πολιτών και ας αφήσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια τύπου επώνυμα και άλλα τέτοια της μητέρας μας. Τώρα, στον έλεγχο με τα φανάρια κυκλοφορίας που αναφερθήκαμε ε, δεν είναι ότι μπορούμε να έχουμε ένα τροχονόμο σε κάθε σταυροδρόμι για να παρακολουθούμε πώς είναι η κυκλοφορία σε όλα τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα. Τώρα, ε, αν η Κομισιόν θεωρήσει ε, ότι μία πρόταση είναι σοβαρή, συγκεντρώνει μία ευρία στήριξη από τους πολίτες, ας μην μπαίνουμε σε τρεις λεπτομέρειες όπως τα ονόματα αυτά που είπατε και διάφορα άλλα τεχνικά, ώστε τα πράγματα, εν περιπτώσει, να κινούν πιο ομαλά και να παρακολουθούμε τις προτάσεις των πολιτών. Ε, αν έχουμε χρόνο, Πρόεδρε, Τώρα είναι τρία χρόνια που συζητούμε αν πρέπει να είναι πόσα, ε, τι αριθμοί πολιτών, πόσες υπογραφές, τι συνθήκες, είναι στη συνθήκη, όλα αυτά είναι σαφή. Συζητούμε αν πρέπει να πάρουμε σοβαρά αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι στη συνθήκη όμως. Τώρα γνωρίζω την ε, τοποθέτηση του κυρίου Κόλμπετ από την αρχή. Καλό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, όμως ο Γιώργη θα πρέπει να βρει μια συμβαστική λύση θα θέλατε να σχολιάσετε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια που άκουσα. Αυτό που θα μπορούσα να είχα πει νωρίτερα, θα το πω όμως τώρα, είναι ότι αν θυμάστε, όταν είχε έρθει εδώ ο αντιπρόεδρος κ. Τίμερμαντς, έθεσα αυτό το ερώτημα, όχι μόνο εγώ και άλλοι. Και είπε τότε ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδρασε ε, εντός ε, των πλαισίων της της ε, νομιμότητας. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν νομικές πτυχές στην πολιτική βούληση. Τώρα, κυρία Κάουφμαν, να σας πω ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κανονικά θα έπρεπε να είναι έτοιμη στο τέλος του μήνα, 31 Μαρτίου, Απριλίου, εκεί. Το που καταλαβαίνω εγώ χωρίς να έχω δει το κείμενο είναι ότι εν μέρη μας περιμένουν να δουν τι θα κάνουμε. Ε, και η έκθεση αυτή θα είναι αρκετά τεχνική και θα εστιάζεται στα γεγονότα. Όμως, κατά τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, στα τέλη δηλαδή του 2015, θα υπάρχει μια μεγαλύτερη έκθεση, η οποία θα είναι λεπτομερέστερη. Υποθέτω, χωρίς να έχω δει τα κριτήρια της ε, Κομισιόν. Τώρα, σχετικά με τα 16χρονα και το δικαίωμα ψήφου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι ενδέχεται κάποια κρατημέλη να έχουν. Και σίγουρα χρειάζεται να συζητηθούν οι λεπτομέρειες, όμως ναι, θα ήταν κάπως περίεργο αν σε κάποια κρατημέλη ψήφιζες από τα 16 και αν σε κάποια άλλα από τα 18. Βέβαια, να το κοιτάξουμε, όπως είπατε τώρα, ε, το πρόγραμμα που είπατε. Ελπίζουμε η έκθεση να συζητηθεί για δεύτερη φορά εδώ και μετά να την ψηφίσουμε το Μάιο ή τον Ιούλιο και ιδανικά να πάει στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή να είναι έτοιμη πριν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα τέλη του 2015. Τώρα, Φυσικά και συμφωνώ με εσάς ότι δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε ένα μέσο το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και όπως είχα πει σε μια κατηδίαν συζήτηση, έτσι γεννιούνται οι ευρωσκεπτικιστές. Ρίτσαρντ, τώρα ναι, ναι, ναι, εσύ με αυτές τις δυσίωνες σκέψεις που κάνεις να αντιπροτείνω κάτι. Δεν αρκεί μόνο να πούμε ότι ναι, είμαι Ευρωπαίος πολίτη, έχω μια καταπληκτική ιδέα, Α κάνουμε κάτι. Όχι, υπάρχουν Υπάρχει μια διαδικασία όπου εσύ εμπλέκεσαι στη διοργάνωση ενός ε, κινήματο ε, μιας πράξη από τη βάση προς τα πάνω και αυτό είναι το θετικό και πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό είναι να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Τώρα εντάξει δεν θα κολλήσουμε στο 1.940.000-980.000 υπογραφές όπως και να έχει. Πιστεύω πως αν πάρουμε στα σοβαρά αυτό το στοιχείο της κινητοποίησης των πολιτών σίγουρα θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος διότι Έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις πως ήταν πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία της καταγραφής και ότι εκεί μετά από την καταγραφή χρειάστηκε αρκετός χρόνος έτσι ώστε να οργανωθεί το πράγμα. Όμως η πρωτοβουλία των πολιτών είναι σίγουρα ένα μέσο που πρέπει να διατηρηθεί, οφείλει να διατηρηθεί και να πω Επίσης και ότι από τη στιγμή που δημιουργείται ένας θεσμός, όπως η πρωτοβουλία των πολιτών, δύσκολα αλλάζει. Διότι διαμορφώνεται ένα μοτίβο εργασίας, το συνηθίζουν οι πολίτες και μετά είναι δύσκολη οποιαδήποτε αλλαγή ενδεχόμενη, η κατάργηση. Και πιστεύω λοιπόν πως προτιμότερο είναι να το αναδιαμορφώσουμε λιγάκι, να το τροποποιήσουμε παρά να ξαναγυρίσουμε στην φάση του σχεδιασμού. Μάλιστα, λέει πρόεδρο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθετε και στι 16 Απριλίου θα έχουμε στην Επιτροπή μια γραπτή έκθεση. Πολύ ωραία, σα ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα περνάμε πάλι στο Ρίτσαρντ. Και στην έκθεσή του σχετικά με τι διαδικασίε και τι πρακτικέ ε, όσον αφορά τι ακροάσει των επιτρόπων να σας υπενθυμίσω ότι σας ζητήσαμε να είστε εισηγητής και μετά σας ζητήσαμε να συντάξετε μία έκθεση και τώρα θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης. Ρίτσαρντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίω έκανα την προηγούμενη, το προηγούμενο έγγραφο εργασίας μου σε μία έκθεση με ένα σχέδιο ψηφίσματος. που περιέχει τα πορίσματα της διαδικασίας ε, αποτίμησης των ακροάσεων των επιτρόπων. Άρα δεν θα υπάρξουν, δεν υπάρχουν εκπλήξεις στο κείμενο αυτό. Αντανακλά πλήρως αυτά τα οποία είχε το εγγραφό εργασία, συζητήθηκε στη διάσκεψη των Πρόεδρων Επιτροπών, ε, σε κάποιες πολιτικές ομάδες κτλ. Για τα περισσότερα θέματα υπάρχει αρκετά ευρεία συνένεση. Κάποιε λεπτομέρειε βεβαίω οι συνάδελφοι μπορεί να θέλουν να τροπολογήσουν ελαφρώς. Αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα σημεία είναι όντως αντικείμενο ευρείας αποδοχής. Συναντήθηκα με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Τίμεμαν την προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε τις απόψεις ε, της Επιτροπής για την έκθεσή μου. Δεν εξέφρασε αντιρρήσεις. Θέλουν να είναι σαφείς οι κανόνες και να εφαρμόζονται ισότιμα για όλους τους ε, υποψηφίους επιτρόπους. Λογικό. Ένα θέμα στο οποίο δεν αναφέρθηκα και το ανέφερε ο κύριος Τίμεμανς είναι το θέμα του γραπτού ερωτηματολογίου που στέλνουμε ε, πριν από την ε, ακρόαση στους επιτρόπους. Κάποιες επιτροπές στέλνουν πέντε σύντομες ερωτήσεις ενώ άλλες στέλνουν πέντε ερωτήσεις ε, που η καθεμία περιέχει 12 υποερωτήσεις. Καμία ομοιογένεια λοιπόν. Λογικό. Ότι πρέπει και αυτό να το δούμε. Δεν το είχα εξετάσει μέχρι τώρα. Οπότε να ακούσω τις απόψεις επ' αυτού μέσω τροπολογιών. Αν χρειάζεται. Αυτά ευχαριστώ. πρώτος ευχαριστώ. Ο Γιώργη Σόπλιν. Ευχαριστώ. Εκ μέρου του σκιώδους μας, Κρίστιαν Πρέντα, ο οποίος ζητά συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να παρευρεθεί, είναι στην Άγκυρα με μια αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ. Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο το οποίο μου έδωσε. Συγχαίρει τον κύριο Κόμπερτ για το θαυμάσιο σχέδιο έκθεσης ιδιαίτερα το ότι ο συγητής έλαβε υπόψη τις συζητήσεις που έγιναν το Δεκέμβριο με βάση το έγγραφο εργασία και ότι τα κυρία πορίσματα είναι στο σχέδιο έκθεση. Για την παράγραφο 1. Ο κ. Πρέντα καλωσορίζει την ιδέα να καθοριστεί μια προθεσμία ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να ανακοινώνουν τα ονόματα υποψηφίων επιτρόπων. Το τελευταίο τμήμα τη παραγράφου όμω αφήνει κάποιο περιθώριο ερμηνεία καλή ιδέα να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα για το πώς να εξελιχθεί κατόπιν η διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο καθορισμός προθεσμίας είναι σημαντικός για μας. Για την παράγραφο 3, για το ΕΛΚ είναι επίσης σημαντικό να κάνει μία αποτίμηση για την ακρόαση Τίμεμανς όπου έγινε παράβαση των κανόνων, του εσωτερικού κανονισμού. Και αυτό αφορά όλες τις ακροάσεις επιτρόπων που έχουν οριζόντιες αρμοδιότητες. Αλλά υπάρχει πρόβλημα και όταν ε, οι ακροάσεις συνδιοργανώνονται από τρεις-τέσσερις επιτροπές, να δούμε πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε λοιπόν. Για την παράγραφο 5, όπως είπα και προηγουμένως, ο κύριος Πρέντα λέει ότι πρέπει να είμαστε σαφείς για τις συνεδριάσεις αποτίμηση των ακροάσεων και η έκθεση διευκρινίζει πολύ την κατάσταση του θέματος αυτού. Όμως στην παράγραφο 5, στο εδάφιο 4, υπό εδάφιο, υπό ε, παύλα 3, λέει «Εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει συνένεση, η αίτηση να γίνει μια μισή ώρα παραπάνω». Είναι το δεύτερο εδάφιο της τέταρτης παύλας ο κύριος Πρέντα θα προτιμούσε να γίνεται αυτό το αίτημα από τη διάσκεψη Πρόεδρου και όχι μόνο από τον Πρόεδρο. Για την παράγραφο 6, πέρα από το θέμα της διαφάνειας και της ε, υψηλής διάδοσης των ε, επιστολών αποτίμησης, θα πρέπει να υπάρχει και εναρμόνιση τους. Παρά την κοινή δομή υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση στον τρόπο σύνταξής των. Κατά την προσωπική του γνώμη, οι ακροάσεις πήγαν πολύ καλά. Είχαν ως αποτέλεσμα μία επιστολή ουδέτερη και διοικητική, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πιο ε, λεπτές οι εκτιμήσεις ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Μάιτε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Η έκθεση του συναδέλφου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει μια συνεισφορά πολύ χρήσιμη και πολύ σημαντική αλλά εγώ δεν θεωρώ τόσο ε, χρήσιμο να μειώσουμε τα ερωτήματα που τίθενται στους ε, υποψηφίους επιτρόπους ακροάσεις. Γιατί ε, αυτή η διαδικασία πολλής ερωτήσεων μας επιτρέπει να βλέπουμε περισσότερα στοιχεία της προσωπικότητας Και μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε εκείνο το οποίο καλούμαστε να αξιολογήσουμε στην ουσία επί τη βάση του κανονισμού. Αυτό αφενός. Αφετέρου θα έλεγα ότι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι σε σχέση με τις ημερομηνίε που γινόντουσαν, που γίνονται αυτές οι ακροάσεις, η πολιτική ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ομάδων ήταν τέτοια που η αξιολόγηση, ψυχολογικός πώς, στο πολιτικό πεδίο, ήταν υποκειμενική, πάντα υπάρχει βεβαίω ένα υποκειμενικό στοιχείο, υπάρχουν συμφωνίε μεταξύ πολιτικών ομάδων, υπάρχει πολιτική ισορροπία, αλλά θα έπρεπε στο μέτρο του δυνατού να προσπαθούμε να αξιολογούμε, μάλλον να κάνουμε μια προσπάθεια προς το αντικειμενικότερο, ώστε αυτοί που να πρέπει να εγκρίνονται να εγκρίνονται και αυτοί που δεν πρέπει να μην εγκρίνονται. Μπορούμε λοιπόν σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές που ε, σχετίζονται με την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων να, βελτιώσουμε τα πράγματα πιστεύω. Τώρα, το ένα ή το άλλο χρονικό σημείο εντός της εβδομάδας ή το αν θα μπορούμε να έχουμε κριτήρια πιο αντικειμενικά και βεβαίως πάνω απ' όλα η ποιότητα που αναζητούμε και μας ζητάει ο κανονισμός να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μέσο εξαιρετικά χρήσιμο και οπωσδήποτε πρέπει να συνεχιστεί να συνεχίσουν να υποβάλλονται οι υποψήφοι επίτροποι σε αυτή τη δοκιμασία προκειμένου να εκπροσωπούν καλύτερα δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο Ρίτσαρτ. Δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό πρέπει να καλύπτεται. Αλλά πάντα επίθετο το θέμα του κατά πόσον ελέγχαμε τις υποσχέσεις που είχαν δώσει οι επίτροποι στις ακροάσεις αυτές. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε ως post ακρόαση ως παρακολούθηση του τι είχε πει ο Επίτροπος, τι δέσμευση είχε αναλάβει. Βεβαίω κάποιες από τι δεσμεύσεις αυτέ μπορεί, να μην, μπορεί να αγνοούν και το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασία της Κομισιόν όπου διαμορφώνεται μετά. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει αυτή η εξακρίβωση, αν θέλετε, η επαλήθευση των υποσχέσεων, των δεσμεύσεων του ή της υποψήφιου, υποψήφιας επιτρόπου. Δεν αισθάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Ε, ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Πολύ χρήσιμα. Και συμφωνώ με πολλά από αυτά. Όχι με όλα, αλλά με πολλά. Σημειώνω ότι η διαδικασία Τίμερμανς μάλλον ήταν κατά των κανόνων. Κατά πόσον τώρα πρέπει να εμείνουμε σε αυτό ή όχι ή απλώς να επικεντρωθούμε στο να έχουμε καλύτερους και σαφέστερους κανόνες για το μέλλον, εγώ αυτό θα προέκρινα. Εμπαστός σίγουρα είχαμε απόκληση. Τώρα διατρέχω τα εδάφια και όχι την σειρά όπως αναφέρθηκαν οι ομιλητές για τον αριθμό των ερωτημάτων 25 αντί για 42 είναι σημαντικό να διαβάσετε το σύνολο του εδαφίου όπου κάθε ερώτηση επιτρέπει άμεσα επόμενη ερώτηση, follow-up ερώτηση στην προηγούμενη. Και επομένω συνολικά έχει κανείς σαφώς περισσότερες από 20 από αυτέ που αναφέρουμε. Υπάρχει απάντηση δηλαδή και μετά μπορεί να ζητηθεί μάλλον χωρίς αυτή τη δυνατότητα δεν υπάρχει μια ε, ζωντανή ακροματική διαδικασία γιατί τότε αλλάζουμε θέμα και κλείνει το προηγούμενο και έτσι αυτή ακριβώς ήταν η προσέγγιση μου στην πρόταση τη δική μου. και ίσως με κάποιον συντανισμό μεταξύ των μελών της Επιτροπής με 25 αρχικά ερωτήματα θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλα τα σημαντικά θέματα που πρέπει τότε θα προετοιμάζαμε ίσως και καλύτερα και από πλευράς μας πρόεδρος θέλει μπλε κάρτα η ε, πρόεδρος για άμεση αντίδραση ε, όχι ακούστε όμως όταν έχουμε 40 ερωτήσεις δίνει σαφές δείγμα ο υποψήφιος είτε απαντήσει είτε δεν απαντήσει των δεσμεύσεων και προθέσεών του ή της. Δηλαδή είτε απαντήσει είτε δεν απαντήσει, επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολύ δεικτικό κάποιες φορές. Okay. Uh, ναι, ναι, εντάξει, δεν θέλω κι εγώ να πω ότι είναι μπλε κάρτα. Υποστηρίζω την ιδέα του Ρίτσαρντ. Γιατί νομίζω ότι οι ακροάσεις πρέπει να επιτρέψουν μια δυνατότητα διαλόγου, όχι ερωτήσει μία μετά την άλλη. Δεν έχει κανείς δυνατότητα να αντιδράσει. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ακριβώς να ρωτάει και μετά να «Ναι, να ρωτήσει μια εναλλαγή απόξεων, ένα πινκ-πονγκ ένας ουσιώδης διάλογος. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο τυπικοί και γραφειοκρατικοί στην εργασία μας. Διότι σε τελευταία ανάλυση λιγότερα αποκομίζουν οι βουλευτές στο τέλος για να μπορέσουν να κρίνουν. Οπότε υποστηρίζω απόλυτα την άποψή σου. Χόμπετ. Ναι, βλέπω υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από αυτού αλλά και από τα προηγούμενα που είπαμε η πλειοψηφία νομίζω ήθελε ακριβώς ε, πολύ περισσότερες δυνατότητες διαλόγου να θέτουμε ερωτήσεις για να γίνονται απαντήσεις. Δεν είναι σκοπός της ακρόασης να μιλήσουν όσο να τον περισσότερο βουλευτές. Είναι να γίνει ουσιαστική διερεύνηση των προθέσεων του υποψηφίου επιτρόπου για το σημείο του ΕΛΚ για την παράγραφο 5 τέταρτη σφαίρα, δεύτερη υποσφαίρα ναι μπορούμε να πούμε με την έγκριση της διάσκεψης των Πρόεδρων και όχι απλώς του Προέδρου αλλά μπορεί να υπάρχει ένα διαδικαστικό πρόγραμμα, πρέπει, πρόβλημα γιατί πρέπει να συνεδριάσει η διάσκεψη των Πρόεδρων και αυτό μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία αλλά δεν είναι θεμελιώδες θέμα μία, ένα συγκεκριμένο πρότυπο επιστολής. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί αυτό να μπει στον εσωτερικό κανονισμό. Μπορούμε να το εξετάσουμε χωρίς υποχρεωτικά να μπει στον εσωτερικό κανονισμό. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα. Την προηγούμενη φορά γίνανε οι ακροάσεις όλες ε, πολύ κοντά η μία στην άλλη γιατί μάθαμε τα ονόματα των επιτρόπων ε, πολύ αργά σε σχέση με την προθεσμία 1η Νοεμβρίου που θέλαμε να σεβαστούμε για πολιτικούς λόγους. Άρα επανερχόμεθα στο πρώτο σημείο, να υπάρχει προθεσμία νωρίτερα ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων. Αυτό θα επέλει μια σειρά προβλήματα στην περαιτέρω μετά διαδικασία αν θα πρέπει να θέσουμε και κριτήρια αποτίμησης ε, της απόδοσής τους. Είναι μια πολιτική αυτή η αποτίμηση. Ο καθένας έχει τα κριτήριά του. Πέρα από αυτά που θα καθορίσουμε ή που καθορίζει η συνθήκη, η ανεξαρτησία, η ικανότητα και δέσμευση υπέρ της Ευρώπη. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα από αυτού σε ένα νομοθετικό κείμενο. Είναι μια πολιτική αποτίμηση. Ναι, ορισμένοι από μια πολιτική ομάδα μπορεί να τείνουν να είναι πιο επικριτικοί για τους υποψηφίους επιτρόπους της άλλης πολιτικής οικογένειας και ορισμένοι μπορεί να υπερασπίζονται αυτούς που είναι από τη δική τους πολιτική οικογένεια. μία ή άλλη είναι αυτά. Ένας επίτροπος για να απορριφθεί τελικά απορρίπτεται μόνο αν υπάρχει ευρεία συνένεση ότι δεν θα τα βγάλει πέρα. Γιατί αν μόνο όλοι ψήφισαν τους δικούς τους υποψηφίους επιτρόπους και κατά όλων των άλλων, δεν θα διοριζόταν κανένας. Γιατί κανένα κόμμα δεν έχει πλειοψηφία. Υπάρχει κάποιο δούνε και λαβίν. Που σε τελευταία ανάλυση έχει καλά αποτελέσματα. Γιατί απορρίπτεται κάποιος αν υπάρχει σχετικά ευρεία απόρριψή του. Τώρα πώς μετά θα ελέγξουμε αν τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Αυτό που έκανε η Υπηρεσία Μελετών του Κοινοβουλίου, που συνέταξε έναν κατάλογο των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι επίτροποι, βοήθησε πολύ. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι επιτροπές αυτό το κατάλογο κατά την τρέχουσα πενταετία και όταν από καιρού καιρό έρχονται ενώπιον των διαφορών επιτροπών οι επίτροποι, αυτό ο κατάλογος θα βοηθούσε να πούν ε, οι συνάδελφοι, μα κύριε επίτροπε, η κυρία, είπατε αυτό στην ακρόασή σα και δεν το κάνετε. Τι το ξεχάσατε και λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν χρειάζεται ε, ένας επιπλέον γύρος ακροάσεων στη μέση της θητείας. Νομίζω ότι πρέπει το κατάλογο αυτό να αξιοποιούμε ε, όποτε ε, προκύπτει δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Και άλλη μπλε κάρτα. Α, μάλιστα. Να σας πω την άποψη των πρασίνων. Καλή έκθεση πιστεύουμε. Και την υποστηρίζουμε τουλάχιστον ε, τα μεγαλύτερα τμήματά τους. Λοιπόν, στο σημείο όμως 5, σφαιρίδιο 4, υποσφαιρίδιο 3. Το τελευταίο. Που λέει αν εξακολουθεί να μην υπάρχει συνένεση, η συντηρητική πλειοψηφία μεταξύ των συντονιστών τότε θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή. Θεωρούμε ότι αν μια πολιτική ομάδα θέλει να υπάρξει ψηφοφορία, θα πρέπει να γίνεται ψηφοφορία. Αυτά πιστεύει η ομάδα μου. Και επίσης θεωρούμε ότι η λέξη συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι αρκετά σαφής στο, για να είναι σε ένα κανόνα. 51% είναι η πλειοψηφία. 50% θα θεωρήσουν ότι είναι συντριπτική πλειοψηφία. Εάν θέλουν να θεωρήσουν ότι 51% είναι συντριπτική πλειοψηφία. Για το σημείο 8. Αυτή, αυτό το παλιό τροπάριο για τον έλεγχο. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πρέπει να ελέγχει τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι και σαφέστερο το 8. Ίσως θα έπρεπε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να μπορεί να δίνει ένα είδος πράσινο φως στους επιτρόπους πριν από την ακρόαση. Τέλος, τέλος, τέλος. Οι κανόνες αυτοί είναι τώρα παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού. Άρα η νομική τους ισχύ δεν είναι παρκώς ρωμαλαία. Μήπως κάποιοι από τους πιο σημαντικούς κανόνες για τις ακροάσεις θα μπορούσαν να περιληφθούν στον εσωτερικό κανονισμό. Στα πλαίσια της διαδικασίας ε, του, της ομάδας εργασίας για τον εσωτερικό κανονισμό. Ε, για να απαντήσω αντίστροφα στις ερωτήσεις σας, το τελευταίο που με ρωτήσατε, ναι, νομικά μιλώντας, το παράρτημα έχει την ίδια νομική ισχύ με το σώμα των κανόνων. Όμως πιστεύω πως θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που προτείνεται για λόγους περισσότερης ε, ορατότητας. Έπειτα, να ξεκαθαρίσω ότι χρειάζεται προσοχή όταν λέμε ότι θέλουμε το πράσινο φως της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων πριν την ακρόαση αυτό δίνει και το δικαίωμα βέτο στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων προτού καν αρχίσουν οι ακροάσεις και πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά τι θα κάνουμε εδώ. Η φυστάμενη διαδικασία, όπως την ερμηνεύσαμε πριν από λίγο, λέει ότι αν η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων βρει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει, αυτό πρέπει να γίνει στα πλαίσια της αξιολόγησης από την Επιτροπή που θα διεξάγει την ακρόαση. Χρειάζεται όμως περισσότερη σκέψη για αυτό το θέμα και περισσότερες προτάσεις από εσάς. Τώρα, η πρώτη σας ερώτηση είναι κάτι που με βρίσκει αντίθετο. Ε, εάν μόνο μία ομάδα επιθυμεί να ψηφίσει, για, ε, επιθυμεί να ψηφίσει σε μία επιτροπή, τότε θα έπρεπε να γίνει η ψηφοφορία. Ε, τότε πιστεύω πως θα καταλήξουμε σε μία κατάσταση όπου αυτό θα επαναλαμβάνεται σε κάθε επιτροπή. Θα υπάρχει μία πολιτική ομάδα η οποία συστηματικά θα επιμένει σε κάθε ε, περίπτωση ακρόαση επιτρόπου, όπως θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία στην ε, επιτροπή. Και αυτό πιστεύω πως ε, δεν είναι καλό για το κοινοβούλιο, διότι μόνο μία ψήφος μέτρα νομικά. Η ψήφος του Κοινοβουλίου στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ψήφος όλου του Κοινοβουλίου για όλη την Επιτροπή. Οι ξεχωριστέ ψηφοφορίες δεν έχουν καμία νομική επίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τον πολιτικό αντίκτυπο των δράσεών μας. Και δεν πρέπει να γίνει ρουτίνα αυτή η ψηφοφορία για τον κάθε επίτροπο, σε κάθε επιτροπή. Γιατί εκεί πέρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις όπου κάπου θα υπάρχουν πλειοψηφίε, κάπου όχι. Εάν διατηρήσουμε την δυνατότητα ψηφοφορίας μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου έχει, έχουν αποφανθεί ότι δεν είναι κατάλληλος ο Επίτροπος, τότε θα μεγιστοποιηθεί και ο πολιτικός ε, αντίκτυπος αυτής της διαδικασίας που είναι πολιτική και όχι νομική. Γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με αυτό που είπατε. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Θα μπορούσατε να μας πείτε και ποιος είστε επίσης. Καλησπέρα σε όλους. Φλέμενς ονομάζομαι. Αντιπρόεδρος της ε, Γενικής ε, Διεύθυνσης για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα ελέγχθησαν και να πω ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε και ο εισηγητής. Δηλαδή, η ίση των διαφορών επιτρόπων στις διάφορες ακροάσεις σε σχέση με τον αριθμό των ερωτήσεων που τους υποβάλλονται και την δομή των ακροάσεων η οποία κατά την τελευταία διαδικασία διέφερε από τις προηγούμενες και πιστεύω πως αυτό απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο από όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρίτσαρντ, θα ήθελες να σχολιάσεις? Όχι. Να πω ότι δεν χρειάζεται να λάβουμε κάποια απόφαση εκτός από μία, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών. Έχουμε προτείνει την 24η Μαρτίου, δηλαδή σε μια εβδομάδα στις 6 το απόγευμα. Θα μπορούσαμε να παρατείνουμε την προθεσμία, έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε ευέλικτοι, όμως ε, πολλές φορές αυτό δεν δείχνεται γιατί χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και ξεχνιόμαστε. Για το καλό σας το λέω. Είμαι ευέλικτο, λέει ο εισηγητή. Μετά μεσολαβεί το Πάσχα. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε μία μόνο εβδομάδα παραπάνω. Παραπάνω από μία μπορούμε να σας δώσουμε. «13 Απριλίου, Δευτέρα 13 Απριλίου, είστε εντάξει με αυτό» «Μάιτε, Μα νομίζω ότι είναι πολύ σύντομη η προθεσμία. Δεν μπορεί να επεκταθεί λιγάκι. Μέχρι τις 13 Απριλίου να επεκταθεί. Ωραία, 13 Απριλίου, πρόεδρος. Ωραία. Παρατείνεται μέχρι τις 13 Απριλίου η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. 18 η ώρα, 6 ώρα το απόγευμα. 13 Απριλίου, 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, ένας συνάδελφος από την Κομισιόν, η Κάρμεν Πράισινγκ, ήθελε να μιλήσει για το θέμα του Γιώργη, αλλά δυστυχώς το ξέχασε. Λυπάμαι, λυπάμαι. Παρακαλώ να διαβιβάσετε στο συνάδελφό σα ε, τη συγγνώμη μου. Το επόμενο θέμα είναι πολύ δύσκολο, γιατί η κατάσταση είναι η εξή. Ο κύριος και ο εισηγητής μας, για το επόμενο θέμα, και το μάθαμε τώρα, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Είναι οι αιτήσει εκθέσει 12-13 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη συνεδρίασή μας ο κύριος Βουγιαντόφσκι έκανε μια εισαγωγή για το θέμα του, αλλά δεν υπήρχε χρόνος για να συνεχιστεί η συζήτηση και αναβλήθηκε μέχρι σήμερα, αλλά σήμερα λείπει. Αν η είναι διατεθειμένη θα ήθελαν να σχολιάσουν και μετά θα συζητήσουν ε, με τον κύριο Γιαντόφσκι για τις τροπολογίες. Αν συμφωνούν οι σκιώδεις, παρά το γεγονός ότι λείπει ο συγκητής, εντάξει. Ωραία, ποιος θα ξεκινήσει. Α, ο Γιώργη. Ναι, ναι. Ωραία, πρώτο το ΕΛΚ. Ο κύριος Πρέντα δεν έχει γυρίσει εδώ και μια μισή ώρα από την Άγκυρα. Να σας διαβάσω λοιπόν το κείμενο που μου έδωσε. Πρώτα απ' όλα συγγνώμη που λείπω. Πολύ θα είχα ευχαριστηθεί την συζήτηση για το σχέδιο γνωμοδότησης για τις εκθέσεις 12-13 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Δυστυχώς δεν μπορώ. Γιατί είμαι στην Τουρκία. Ευχαριστώ τον κύριο Γιαντόφσκι για τη θαυμάσια εργασία του για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Το κείμενο το οποίο συνέταξε τονίζει βασικά σημεία τη εφαρμογή, τη αρχή τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Όπω και ο κύριο Γιαντόφσκι θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη σημασία τη εξάντε εξακρίβωση για τι προτάσει τη Κομισιόν για το εάν και κατά πόσο σέβονται την επικουρικότητα και αναλογικότητα και θεωρώ ότι οι ιδεολογημένε γνώμε των Εθνικών Κοινοβουλίων και ο αυξανόμενο αριθμό του είναι θετική τάση, ελπίζω να συνεχιστεί. Επίσης, η διαφορετικότητα των κριτηρίων που χρησιμοποιούν τα Εθνικά Κοινοβούλια για να αποτιμήσουν το σεβασμό της επικουρικότητα και της αναλογικότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σοβαρό θέμα, γιατί ορισμένες φορές ε, δεν γίνονται αποτιμήσει με βάση τα ίδια κριτήρια. Θα έπρεπε λοιπόν να συζητήσουμε για τα κριτήρια και τι μεθόδου αποτίμηση των αρχών τη αναλογικότητα και τη επικουρικότητα. Επιπλέον, θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί. Τα εθνικά κοινοβούλια που έχουν ήδη σημαντική πείρα στην αποτίμηση τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Οπωσδήποτε πρέπει λοιπόν να συμμετάσχουν. Θα ήθελε η έκθεση να τονίζει τον αυξανόμενο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο εκθέσεις αναφέρουν ακριβώς πόσο θετικά αποτιμούν αυτό το ρόλο. Τέλος θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε περαιτέρω ότι ενθαρρύνουμε τα τοπικά και περιφερειακά κοινοβούλια, όχι μόνο τα εθνικά, να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό πιστεύω ότι ε, είναι σύμφωνο με τις αρχές ε, ε, συμμετοχής όλων που εισάγει η αρχή της, που εισάγει η συνθήκη της Λισαβόνας. Η Μερθέδας Βρέσο για τους σοσιαλιστές. Κοιτάξτε, εγώ ε, είχα ένα σημείωμα που δεν θα διαβάσω, αλλά... Αλλά... Διακόπτει μου, γιατί... Μπορώ όμως να σας το υποβάλω ώστε ο εισηγητής να έχει ένα σημείωμα που να μπορεί να το λάβει υπόψη του για τις τροπολογίες. Τώρα συμφωνώ με τον κύριο Σόπλινγκ, δηλαδή στην ουσία με τον κύριο Πρέντα και την παρατήρηση ότι είναι σημαντικό καταρχάς ότι πρέπει να σεβόμαστε και την επικουρικότητα αλλά και την αναλογικότητα γιατί πολύ συχνά το θέμα άπτεται της αναλογικότητας και ο έλεγχος της πρέπει να εντάσσεται, να ενσωματώνεται στον έλεγχο της επικουρικότητας. Είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια μιας επιτροπής όπως η δική μας. δεν κοιτάζει μόνο το γράμμα του κανόνα αλλά και το πνεύμα. και είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μα και τις παρατηρήσεις που υπάρχουν από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Συμφωνώ και με κάποιε από τις επικρίσεις, δηλαδή η πολύ περιορισμένη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή τη συμμετοχή και θα πρέπει μέσω της συμμετοχής τους να αυξήσουμε την νομιμότητα αλλά και την πληρότητα της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτή η συμμετοχή που είναι περιορισμένη παρότι έχει αυξηθεί κατά τη εξηγείται μέσω των προθεσμιών που είναι αρκετά ασθενές. Οκτώ εβδομάδες για τα εθνικά κοινοβούλια είναι πάρα πολύ μικρό διάστημα διότι πάντοτε υπάρχει πέρασμα μεταξύ επιτροπής, ολομελία κτλ. Οκτώ εβδομάδες είναι πολύ στενή η προθεσμία. Υπάρχουν και ολομέλειες, υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν ημερομηνίε που παρεμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει. Ίσως θα έπρεπε να το ξαναδούμε δηλαδή, το διάστημα αυτό. Επίσης, θεωρώ, συμφωνώ, ότι πρέπει να ενισχύσουμε το δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων και θα έλεγα θα προσέθετα και των περιφερειακών ή τοπικών κοινοβουλίων γιατί και αυτά έχουν ρόλο μέσω των εθνικών του κοινοβουλίου διότι μπορούν να θέτουν ένα θέμα παραβίασης επικορικότητας και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την προθεσμία των 8 εβδομάδων. Γιατί εφόσον έχει δικαίωμα ένα τοπικό κοινοβούλιο να υπογραμμίσει μια μη συμμόρφωση επικορικότητας ή αναλογικότητας προς το Εθνικό Κεντρικό Κοινοβούλιο και μετά το Εθνικό Κοινοβούλιο πρέπει να το επισημάνει το ίδιο σε εμάς οι οκτώ εβδομάδες είναι απολύτως ανεπαρκείς. Και για να ολοκληρώσω θεωρώ ότι θα έπρεπε να προτείνουμε στην Κομισιόν να προτείνει κάποιε κατευθυντήριε γραμμές προκειμένου να βελτιωθεί η όλη αυτή η διαδικασία και να ενσωματωθούν καλύτερα σε αυτήν τα εθνικά και τοπικά κοινοβούλια. Και θα πήγαινα ένα βήμα πιο πέρα από τον εισηγητή, προσθέτοντας ότι θα ήταν ενδεχομένω ενδιαφέρον στην ε, γνωμότηση αυτή να προσθέσουμε μια μικρή φράση για την ανάγκη συσχετισμού, πιο εντατικού συσχετισμού με άλλους θεσμικούς φορείς, εγγυητές επικορικότητας, υπάρχει η Επιτροπή των Περιφερειών, αναφέρω, που σύμφωνα με τη συνθήκη είναι ένας από τους θεματοφύλακες και μέσω αυτής και μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπως έλεγα, τα τοπικά και περιφερειακά. Ανάλογα, εν πάση περιπτώσει, με την ονοματολογία που τους δίδεται στη χώρα τους. Αλλά ε, και ως προς αυτό θα έπρεπε ίσως να προσθέτουμε κάτι, δεν ξέρω αν ο εισηγητής ο ίδιος θα μπορούσε να το κάνει, Ιδάλλως θα μπορούσαμε να υποβάλουμε κάποια πρώτε τροπολογίες. Επίσης θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάτι σαν πράσινη κάρτα των βουλευτών ώστε να δίδεται όχι τυπικό δικαίωμα πρωτοβουλία στα εθνικά κοινοβούλια, αλλά η δυνατότητα υποβολής ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> θεμάτων, θεματικών επί των οποίων θα επιθυμούσαν να υπάρξει μια παρέμβαση πρωτοβουλία της Κομισιόν. Προτάσεις δηλαδή, θεμάτων που θα άξιζε να εξεταστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Αυτά. Κατά τα άλλα, η γνωμοδότηση στο σύνολό της είναι καλή και θα περιμένουμε βεβαίως και τις ενδεχόμενες άλλες τροπολογίες για να τοποθετηθούμε πλήρως. Τώρα, για τους φιλελεύθερους, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει εκ μέρους του συναδέλφου που λείπει. Ναι, ο κύριος Γκέρεν δεν είναι εδώ, αλλά στην ουσία συμφωνούμε με τη γενική κατεύθυνση. Η κυρία Μπρέσιο τονίζει αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η άξια αυτού του δημοσίου διαλόγου η αναζήτηση μέσων, εργαλείων, μέσω των οποίων και τα εθνικά κοινοβούλια να ενέχονται στη διαδικασία, να συμμετέχουν πιο ενεργώς Ε, σχετικά με θεματικές που θα μπορούσαν να προβληματίζουν να είναι ακαθόδη σημεία για τα εθνικά κοινοβούλια. Και το θέμα της παράσινης κάρτας όπως και της κίτρινης θα το συζητήσουμε. Αλλά εν πάση εδώ συνολικά ε, η πρόταση είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Χρυσόγενος για την ΚΟΕ. I feel αισθάνομαι πως πρέπει να γίνει αναφορά στο θέμα της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Σχετικά με την εφαρμογή του των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής για τα κράτη-μέλη που έχουν μεγάλα ε, ελλείμματα. Είναι ένα θέμα στα πλαίσια του γενικότερου θέματος της εφαρμογής του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων για αυτά τα προγράμματα και τις πράξεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Επίσης, σχετικά με τις αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ για το ίδιο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνει αναφορά στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Μαξ Άντερσον για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πιστεύω εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί η διαδικασία της κίτρινης κάρτας ε, στον έλεγχο της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Χρειάζεται να ενισχυθούν τα εθνικά κοινοβούλια και να συμπεριληφθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχύσουμε την Ευρώπη. Αυτή η πρόταση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και τη στηρίζουμε. δεν μπορούμε να έχουμε κάποια αντίδραση από τον εισηγητή και ελπίζω η βοηθοί του να του μεταφέρουν τα σχόλιά μας. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε να μιλήσει. Όχι. Να προτείνω λοιπόν καταληκτική ημερομηνία για υποβολή τροπολογιών να είναι σύντομη διότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ετροπολογίες της 16 Απριλίου. Προτείνω λοιπόν 23 Μαρτίου, σε μια εβδομάδα να είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών. Είναι Δευτέρα. Όχι. Δεν γίνεται Δευτέρα μεσημέρι, άρα Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα. 23 Μαρτίου. ...23 Μαρτίου λοιπόν στις 6 το απόγευμα ε, προθεσμία υποβολή τροπολογιών και έπειτα 16 Απριλίου θα συζητηθούν οι τροπολογίες μαζί με τον εισηγητή. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Πιστεύω πως εδώ έχουμε τουλάχιστον τους κοιόδους φυγητές. Είναι μια γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τον κανονισμό για το ταμείο αυτό. Εγώ προσωπικά ορίστηκα εισηγήτρια για το ΕΛΚ και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την προσέγγισή μου σχετικά με την γνωμοδότηση αυτή. Καταρχάς, Πιστεύω πως ε, όταν κάνουμε γραμμοδοτήσεις πρέπει να μένουμε εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων μας. Και πρέπει λοιπόν να δείξουμε κάποια συγκράτηση. Έπειτα. αυτό που με καθοδήγησε στην ε, σύνταξη της νομοδότησης είναι ότι έχουμε ένα μέσο άνευ προηγουμένου το οποίο από τη μία αποσκοπεί στο να δώσει μεγαλύτερη όθηση στις επενδύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να δώσει κίνητρο για επενδύσεις στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας έναν πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό εγγυήσεων που αυτό δημιουργεί μία νέα μορφή διοργανικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΤΕ και εξωτερικών φορέων, τραπεζών, με τα κράτη-μέλη και με ιδιωτικού επενδυτές. Πιστεύω πως αυτός ο μηχανισμός δημιουργεί κάτι πραγματικά ευρωπαϊκό, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά μέσα που είχαμε μέχρι τώρα. Εδώ δεν υπάρχουν πλέον τοπικά και περιφερειακά επίπεδα, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο λαμβάνονται και οι αποφάσεις, υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, τίθενται οι προτεραιότητες ε, της ε, πολιτικής και ο συντονισμός αυτών, καθώς και οι προτεραιότητες για συγκεκριμένα έργα. Και αυτή λοιπόν η διοργανική διάσταση δημιουργεί και πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για ένα σύστημα διάφανο, υπεύθυνο και ανοιχτό στη λογοδοσία. Και η δική μας Επιτροπή έχει να συνεισφέρει πολλά στην ε, δημιουργία αυτού του μέσου ιδιαίτερα στον ε, τομέα διασφάλισης της ε, διαφάνειας και της ε, λογοδοσίας. Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην δομή, στη διοικητική δομή και στην αποφυγή πολιτικοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται στα πλαίσια του μέσου αυτού. Επίσης, ασχολήθηκα με το θέμα της διαφάνειας στην επιλογή των εμπειρογνωμόνων, στην επιλογή των κριτηρίων, στην επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, διότι είναι ύψης της σημασίας, πιστεύω. Επίσης, τονίζω και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υποβολή εκθέσεων. Πιστεύω πως παρότι σε άλλες επιτροπές θα δούμε άλλες τροπολογίες, σε άλλες ε, κατευθύνσεις, εδώ εμείς δεν πρέπει να επιμείνουμε στον ρόλο του Κοινοβουλίου εκ των προτέρων στη διαδικασία. Θα προτιμούσα λοιπόν να δω ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα παίζει ρόλο εκ των υστέρων, δηλαδή με διαδικασίες ελέγχου. πιστεύω πως ο έλεγχος που θα ασκήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις, σε αυτές τις εγγύησεις που θα δοθούν, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται υπευθυνότητα στον έλεγχο. Επίσης, έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες οι οποίες κατά τη γνώμη μου θα βελτιώσουν την ισορροπία αυτών που ήδη συμπεριλαμβάνοντας τον κανονισμό και αυτών που πρόκειται να συμπεριληφθούν. Και πιστεύω επίσης πως ο κανονισμός πρέπει να διευθετήσει όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα. Φυσικά και η ΕΤΕ θα χρειαστεί να συμφωνήσει σε λεπτομέρειε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμω όπω είπα στοχεύω στην ε, πληρέστερη και καλύτερη βελτίωση της λειτουργίας όλου του συστήματος. Τώρα, κάτι άλλο θα ήθελα να σας πω σήμερα σχετικά με τις τροπολογίες μου. Όπως γνωρίζετε, θα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός ευελιξίας στα πλαίσια του ε, Συμφωνού Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στις ε, διατάξεις του ΕΦΣΥ, αλλά η Eurostat έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα συνεισφέρει πολύ σημαντικά με την παροχή στατιστικών στοιχείων. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεισφορά της Eurostat προτού ολοκληρωθεί νομικά το θέμα αυτό. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος μετά την έγκριση του κανονισμού να προκύψει η Eurostat με μεθοδολογία, με διάφορα στοιχεία και να ανακαλύψουμε ότι δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, δεν τηρούνται κάποια κριτήρια. Και ενώ ε, εκείνους που θα είναι οι χρήστες του μηχανισμού αυτοευελιξίας Αυτές ε, λοιπόν τις ανησυχίες μου και τις σκέψεις μου τις διατύπωσα με μορφή τροπολογιών στη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Θα ακούσουμε τώρα και τους σκιώδεις εισηγητές Νομίζω πως η Μερσέντες Μπρέσο θα εκπροσωπήσει τους σοσιαλιστές και ο κύριος Χρυσόγονος ε, την ΚΟΕ. Δεν νομίζω πως έχουμε άλλες πολιτικές ομάδες παρούσες. Όμως, αν κάποιος επιθυμεί να τοποθετηθεί και να οριστεί από μόνος τους και ο δεσηγητής, παρακαλώ να το κάνει. Και τώρα θα ήθελα να αρχίσει λοιπόν η συζήτηση με την Mercedes πρώτη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι <clears throat> συμφωνώ με την τοποθέτησή σας ότι οι τροπολογίες μας πρέπει να είναι συνεπείς προς τη λειτουργία, προς την εντολή της Επιτροπής μας και να μην μπαίνουμε στην ουσία των τροπολογιών αρμοδιότητας άλλων επιτροπών. Άρα, πρώτη παρατήρηση η εξής. Αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που επιχειρείται να δοθεί μια σαφήνεια, μια σαφέστερη εξήγηση του Growth Pact που είναι και ένα συμπλήρωμα και θεσμικό της όλης αρχιεκτονικής. Και η δεύτερη παρατήρηση προκύπτει από την πρώτη. φαίνεται προφανέ ότι προσπαθώντας να προωθήσει την ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες διότι δεν έχει μέσα που να τις επιτρέπουν να παρέμβει με θεσμικό τρόπο επί μιας τόσο σημαντικής κρίσης σχετικά με τη δυνατότητα επενδύσεων που είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική μεγέθυνση η ανάπτυξη. Γιατί χωρίς όθηση, υποστήριξη των επενδύσεων δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση και μεταξύ των επενδύσεων χρειάζονται και δημόσιες επενδύσεις. Και επομένως ίσως θα ήταν χρήσιμο να θυμίσουμε ότι η θεματική που την αναφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας των ιδίων πόρων δεν μπορεί πλέον να το παρακάμπτουμε. Γιατί αυτό που φαίνεται προφανές ε, στο σχέδιο Juncker είναι ότι είναι ένας προϋπολογισμός απολύτως ακαμπτός που δεν επιτρέπει την επέκτασή του ούτε μέσω νέων πιστώσεων ούτε με νέων εσόδων ούτε αφήνοντας κανένα άλλο παράθυρο ή δυνατότητα σχετικά με μια παράλληλη εν περιπτώσει διαπραγμάτευση που διεξάγεται για το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Και οι ίδιοι πόροι με δύο τρόπους μπορούν να υφίστανται Δηλαδή είτε με τα άμεσα έσοδα που έχουμε είτε με άλλου είδους εξουσιοδοτήσεις κρατήσεων και επόμενος πρέπει να φτιάξουμε ένα ολόκληρο κάστρο από από τα για να μπορέσουμε να φτάσουμε τελικά στην καρδιά στο θεμελιώδες σημείο του, του, του πλαισίου των συμφωνιών που ενδεχομένως θα πρέπει και αυτό τελικά να ενταχθεί στη συνθήκη. Και είναι θεσμικό το θέμα. Δηλαδή είμαστε εξαναγκασμένοι να διερευνούμε ένα, ένα πλαίσιο, πώς να το πω, όχι απόλυτα θεμητό, εξέβρεση σπόρων από το Horizon, που είχε ήδη αποφασιστεί, και να έχουμε μια περιπλοκότατη και ε, επικίνδυνη δομή, τραπουλόχαρτα που έλεγα πριν, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να επανακινήσουμε στην Ευρώπη την οικονομική μεγέθυνση. Δηλαδή υπάρχουν πολύ σημαντικά σημεία και συμφωνώ μαζί σας σε όλα αυτά που είπατε για τη διαφάνεια, για την ε, ex post επαλήθευση, για την υποβολή στο κοινοβούλιο κτλ. Και βεβαίως θα τα συζητήσουμε αυτά συζητώντα τι τροπολογίε. Αλλά υπάρχει το πρωταρχικό ζήτημα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ευελιξία μέσα σε αυτήν την κρίση διότι δεν διότι έχουμε πρόβλημα ιδίων πόρων και εξαναγκαζόμαστε σε μια επιχείρηση χρηματοπιστωτικής ε, μηχανικής καινοτομίας αλλά ε, εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικούς πόρους αυτούς που υφίστανται, αλλά ε, δεν έχουμε, δεν έχουμε αρμοδιότητα να εξεύρουμε ίδιους πόρους. Παρότι, παραλαμβάνω, αυτό αναγράφεται στη συνθήκη και επομένως δεν είναι εκτός της εντολής των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα των ιδίων πόρων είναι ολοένα και πιο επίγον, ιδιαίτερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, που σαν συνομοθέτης επί του προϋπολογισμού, αν δεν μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα ως προς τα έσοδα, δεν ξέρω σε τι άλλο επηρεάζει. Πρόκειται λοιπόν για θεσμικό θέμα, θεσμικό. Και όχι απλώς, μάλιστα όχι απλώς. Δεν είναι καθόλου θέμα των επιτροπών των επιμέρους. Και πολύ τελευταίο, ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα, Τελευταία παρατήρηση, πάντα μιλώντα υπό την οπτική γωνία τη θεσμική. Πρέπει να θυμίσουμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η δέσμη επενδύσεων θα πρέπει να σέβεται μία από τις βασικότερες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη σύγκληση της εδαφικής και οικονομικής. Γιατί είναι θεμελιώδες με την κυριολεκτική έννοια σημείο αρχή και δεν μπορεί να παραβιάζεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγονος. Α, συγγνώμη. Η Μάιτε ήταν πριν και μετά ο κύριος Α, όχι, όχι, η Γκου είναι μεγαλύτερη έτσι, δεν είναι. Καλώς, καλώς, καλώς, καλώς. Οι κυρίες προηγούνται. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ συνοπτικά. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο σκιώδης από την ομάδα μας αλλά εγώ ε, θεωρώ ότι τα επιχειρήματα που παρουσιάσατε είναι πολύ καλά και ιδιαίτερος αυτό που είπε η κυρία Μπρέσο. Χρειαζόμαστε επιγόντως αυτούς τους μηχανισμούς, πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να μπορέσουμε να τα δούμε. Πρέπει να έχουμε τους επαρκείς ίδιους πόρους, δυνατότητα ε, χρέωσης, όλα αυτά είναι θεμελιώδη αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και για να αποφύγουμε τόσο περίπλοκους μηχανισμούς όπως αυτούς που είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Χρυσόγονος. Φυσικά δεν είμαστε εμείς κύριος Αλμόδη για αυτό το θέμα. Συμφωνώ κυρία Πρόεδρε ότι πρέπει να τονίσουμε περαιτέρω τη διαφάνεια, τη δημοκρατική λογοδοσία την ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και την καταπολέμηση απατών κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Όμως δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο ότι θα προχωρήσει αυτή η ιδέα. Αμφίβολο εάν και κατά πόσο θα πιάσουμε τόσους πολλούς ιδιωτικούς επενδυτές, τόσες πολλές ειδικές επενδύσεις με τόσο λίγο δημόσιο χρήμα. Πρόεδρος. Α, και πράσινη. Ο Μαξ Άντερσον. Δεν νομίζω ότι οι πράσινοι έχουν αποφασίσει ποιος θα είναι ο σκιώδης. Τους διάβασα την έκθεση, τη συζητήσαμε και γενικά θεωρούμε ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές είναι πολύ καλές και υποστηρίζουμε τη γενική προσέγγιση του εισηγητή. Και η Μπάρμπαρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω, να προσθέσω δύο πράγματα σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, Χρυσόγωνος με τον οποίο συμφωνώ. πέρα από την ε, ανεξαρτησία του, του ταμείου αυτού, των πόρων αυτών, θα πρέπει να έχει και κατάλληλη νομική προσωπικότητα και να έχει πιο μόνιμη δομή και σύσταση. Και θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής εντολή σχετικά και διαφοροποίηση των, δημοσίων πόρων και διαχωρισμός τους από, το, από, το, από τους ιδιωτικούς. σημαντικοί οικονομολόγοι, όχι μόνο ο κύριος Βαρουφάκης, ο Υπουργός, ο Ρίτσαρντ Κό, ο κύριος Ματζουκάτο, είπαν ότι η ελπίδα που δημιουργούν οι δημόσιοι πόροι ε, που θα μπορούσαν δηλαδή να ε, ε, κινητοποιήσουν αυτά τα άνω των 300 δις είναι περιορισμένα μέχρι και αστεία. Οι δημόσιοι, οι ήδη πόροι είναι θεμελιώδες ζήτημα και κεντρική σημασία, αλλά πάνω απ' όλα απευθύνουμε στην κυρία Μπρέσο αυτή τη στιγμή είναι ιδεολογικό το βασικό μας πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση που πρέπει να γίνει στο τι είναι δημόσιο και τι είναι ιδιωτικό. Εάν η στόχευσή μας είναι αποκλειστικά στο ιδιωτικό, δεν πρόκειται να καταφέρουμε και πολλά πράγματα. Και σύμφωνα με τον κύριο Κο, τον ε, Ιάπωνα οικονομολόγο, η μεγάλη ύφεση της Ιαπωνίας εξηγείται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο ότι στηρίχθηκαν ακριβώς στους ιδιωτικούς πόρους οι οποίοι δεν κατάφεραν να βρουν διέξοδο από τον κύκλο αυτόν, τον φαύλο κύκλο στον οποίο είχαν μπει. Η κυρία Μπρέσο ήθελε να απαντήσει. Ναι, Πρόεδρε, τουλάχιστον για να εξασφαλίσω ότι ήταν σαφή αυτά που είπα. Δεν συμφωνώ με τη συνάδελφο Σπινέλη ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, λέει η κυρία Μπρέσο. Διότι έχουμε κεφάλαια, έχουμε πόρους που δεν επενδύονται αυτή τη στιγμή. Τα 21 δισεκατομμύρια ακριβώς χρησιμεύουν, αν τα καταφέρουν, εν πάση περιπτώσει, να κινητοποιήσουν τα ιδιωτικά κεφάλαια. Και άρα είναι χρήσιμο το πλάνο, το σχέδιο Juncker. Όμως, είναι σαφές ότι αυτό έχει διατυπωθεί έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους πέραν του πολιετούς υφισταμένου δημοσιονομικού πλαισίου από το οποίο δεν μπορούμε να κονηθούμε ένα, μία σπιθαμή. Και η Κομισιόν και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό εγώ έλεγα ότι πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει συνθήκης πρέπει να έχει ίδιους πόρους και πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιθώριο ευελιξία στη λήψη απόφαση για τον προϋπολογισμό. Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε σημαντικές δημόσιες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και από εκεί πέρα το σύμφωνο σταθερότητας και το πόσο μπλοκάρει τις επενδύσεις για την πλειοψηφία των χωρών, γιατί είναι πολλές οι χώρες που δεν έχουν δημοσιονομικά περιθώρια και επομένως οδηγούμαστε στην ανυπαρξία δημοσίων επενδύσεων. Για τον πολλαπλασιαστή, εγώ έχω άλλες πληροφορίες. Ο δικός μας χρηματοπιστωτικός φορέας λέει ότι μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερο περιθώριο. Αν τραβάει η βάρκα γιατί τότε μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερος, ε, μεγαλύτερα μεγέθη, μεγαλύτερους αριθμούς, γιατί είχαμε περιπτώσεις από τις πληροφορίες, έμπασε τόση τις επίσημες πληροφορίες ε, από τους φορείς που πραγματικά παρακολούθησαν αυτά τα πράγματα τεχνικά, δύναται αυτό. Όμως, όμως, αντιμετωπίζουμε αδυναμία ανυπαρξία δυνατότητος κινητοποίησης πρόσθετων ίδιων πόρων. Και γι' αυτό εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα θεσμικό πρόβλημα για τις δημόσιες επενδύσεις αυτού του είδους. Δεν ξέρω αν... Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλα σχόλια. Άρα ένα-δύο ακόμα σχόλια επί της ε, των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σχέδιο μετησεων Juncker. Παρά τις ε, δυσκολίες ε, υπολογισμού, της ρευστότητος κτλ, τα τεχνικά ζητήματα και τα όσα έχουμε στη διάθεσή μας που είναι περιορισμένα ποσά που προέρχονται από τον προϋπολογισμό ως εγγύησης επί τη βάση υψηλής μοχλεύσεως Τέλος πάντων, είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να λάβουμε υπόψη μας ως δυνατότητα συνδυασμού δημοσίων και ιδιωτικών πόρων ώστε οι ιδιωτικές επενδύσεις να παραμείνουν στην Ευρώπη διότι βλέπουμε και πολλές επενδύσεις να φεύγουν και να πηγαίνουν σε χρηματοπιστωτικές αγορές αλλού στον κόσμο. Επομένως πρέπει η, Ευρώπη ε, να καταστεί ελκυστική για διάφορους επενδυτές. Συνταξιωτικά ταμεία μεταξύ άλλων. δεν ξέρω αν κάτι από όλα αυτά θα μπορέσει να αναβαθμίσει αυτόματα <laughs> τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Είναι δύσκολο να το πει κανεί, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή από το να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα που θα κινητοποιήσει τα, την ιδιωτική χρηματοδότηση προς έργα που ναι, θα μπορέσουν να αποφέρουν αλλά θα πρέπει και να εξυγχρονίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία, να την καταστήσουν ανταγωνιστικότερη, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης που δεν θα χαθούν την επόμενη μέρα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις και ζητήματα που μπορεί αυτό το σχέδιο να καλύψει και να επιλύσει, εν μέρη τουλάχιστον και επειδή διάφοροι έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές ε, προϋπολογισμού, σε συναντήσεις ε, με εκπροσώπους ε, της βιομηχανίας και πρέπει να δημιουργήσουμε και το κλίμα εντός του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αυτές οι, οι επενδύσεις δεν μπορούμε παρά ρεαλιστικά να πούμε ότι δεν θα τα λύσουμε όλα για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει θα χρειαστεί χρόνο, όπως βλέπουμε. Συμφωνώ δηλαδή με όσου εκφράζουν αμφιβολίες και μιλούν για πρόκληση, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα αυτή. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη γνωμοδότηση τη Επιτροπής μας και πρέπει να δούμε τι είναι προσθετημένη αξία και τι όχι. Και μάλιστα πρέπει να το κάνουμε γρήγορα αυτό. Γιατί από την αρχή είχαμε ένα πρόβλημα προθεσμία. Η θέση του Συμβουλίου είναι ήδη επιτάπητος. Η τελική προθεσμία λοιπόν για το σκιώδης είναι 25 Μαρτίου το μεσημέρι και μετά μάλλον θα έχουμε δύο ημέρες περίπου για συμβαστικές. Γιατί μετά θα έχουμε το, τη διακοπή για τον Πάσχα. 25 λοιπόν. 25 λέει η πρόεδρος. 25 Μαρτίου το μεσημέρι. Και μετά ψήφος στην Επιτροπή 16 Απριλίου γιατί στην ε, προϋπολογισμού είναι ήδη 20 η ψήφος. Θα πρέπει όλα αυτά δηλαδή να συντονιστούν. Άρα μεταξύ 25 ε, Μαρτίου και αρχής Απριλίου τέλος πάντων. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ε, δεν θα είμαστε εδώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα έχουμε φύγει. Τέλος πάντων θα είμαστε σε επαφή και θα το δούμε για να μπορέσει να ληφθεί υπόψη. Και με αυτό να κλείσω αυτό το σημείο. Δεν έχω και διάφορα. Επόμενη συνάντηση είναι 16 ε, Απριλίου, πλήρης ημέρα, πρωί για απόγευμα. Αυτά, πέρα της συνεδρίασης.